Thank Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ καλή αρχή, κυρία Υποψήφια Επίτροπε, για την αρχική σας δήλωση. Τώρα θα ακούσουμε τους ομιλητές ε, εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων. Από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ο κύριος Λεβαντόφσκι, έχετε το λόγο. Κυρία Υποψήφια Επιτροπέ, εδώ είμαι. Χρειαζόμαστε πολύ περισσότερες επενδύσεις στην Ευρώπη. Πέρσι είχαμε 15% λιγότερες επενδύσεις από το 2007 και είναι εύκολο να το λέμε έτσι μία εποδός. Χρειαζόμαστε επενδύσεις για ανάπτυξη και δουλειές, αλλά χρειάζεται και χρηματοδότηση και εδώ πέρα ακριβώς υπάρχει το χάσμα μεταξύ λόγων και πραγματικότητας, ειδικά της πραγματικότητας που ζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί στη χώρα σας υπάρχει πρόβλημα με τη ρευστότητα, ειδικά με τις επιχειρήσεις που δεν έχουν ακριβώς πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Από την εμπειρία σας στην Πολωνία, ποια είναι τα πιο ε, υποσχόμενα εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα γιατί εδώ η αγορά αποτυγχάνει. Και όταν μιλάτε με, τις, ε, με τους επιχειρηματίες τι προτιμάνε, επιχορηγήσεις, ε, δάνεια, χρηματοδότηση άλλου είδους. Ευχαριστώ. να σας πω πως ε, πρώτα απ' όλα μετά από 7 χρόνια εμπειρία το συμπέρασμα μου είναι πως δεν υπάρχει έλλειψη χρημάτων. Είναι το να εξοδεύονται τα λεφτά σωστά. Αυτό είναι το ζήτημα. Για να αποδίδουν ακριβώς ε, τη μεγαλύτερη δυνατή προστιθέμενη αξία. γιατί προφανώς υπάρχουν ε, πολλά μέσα διαθέσιμα στο επίπεδο των κρατομελών και της ε, Κομισιόν. Στο δικό μου χαρτοφυλάκιο υπάρχει το πρόγραμμα COSME που ανέφερα ήδη και στο επίπεδο των ε, κρατών μελών υπάρχει και η περιφερειακή πολιτική. Οπωσδήποτε θα αντλήσω από την ε, προηγούμενη εμπειρία μου, αλλά νομίζω πως ε, μπορούμε να πούμε ότι όταν ξοδεύονται σωστά τα κονδύλια της περιφερειακής πολιτικής είναι πολύ αποτελεσματικά και υπάρχει και κάποια μόχλευση από την ε, χρήση τους. Στη χώρα μου το είδαμε αυτό το φαινόμενο Όσον αφορά τώρα την διάκριση μεταξύ διαφορετικών τρόπων στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, να πω το εξής. πρέπει να αναζητήσουμε κάποια μέσα με αμοιβαιότητα που θα μας οδηγήσουν σε μεγαλύτερη μόχλευση που αποτελούν και εγγύησει για όλο το πακέτο αυτό. Παραδείγματο χάρη το κεφάλαιο κινδύνου, τα ε, μέσα τα οποία οδηγούν σε εγγύησει πιστώσεων, αλλά πέραν αυτών θα ήθελα να λάβει υπόψη μια εμπειρία. Πρέπει να σας διακόψω, λέει ο πρόεδρος, έχουν περάσει 10 δευτερόλεπτα, πρέπει να τηρείτε τους κανόνες μας. Μία πρόταση μονάχα μπορείτε να προσθέσετε, αλλά μόνο μία. μία μονάχα φράση. Πολλές φορές λίγα χρήματα για τις επιχειρήσεις οι οποίες ξεκινούν μπορεί να έχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα. Είναι μέσα λοιπόν τα οποία μπορούν να δώσουν τεράστια αποτελέσματα και σε τρία ή τέσσερα χρόνια εξασφαλίζουν ότι μια μικρή επιχείρηση μπορεί να αρχίσει να προσλαμβάνει ε, εργαζομένους. Κυρία Φαν Μπρέμπτ από τη Σοσιαλιστική Ομάδα. Um, <laughs> I'm here. Εδώ είμαι, εδώ είμαι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή αρχική σας δήλωση, αν και πρέπει να πω πως οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες εμείς δεν θεωρούμε πως χρειαζόμαστε πιο φιλελεύθερη Ευρώπη. Χρειαζόμαστε μια Ευρώπη που επενδύει πολύ περισσότερο. Και υπ' αυτή την έννοια μας υποσχέθηκε ο Σαν Κλοντ Γιούνκερ πως θα διαθέσει 300 δισεκατομμύρια για επενδύσεις στην Ένωση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Μιλήσατε για την εκβιομηχάνηση, σημαντικό αυτό. Θα ανασκευάσω κάπως αυτό το οποίο είπατε. Εγώ θα έλεγα πως χρειαζόμαστε εκβιομηχάνηση, αλλά αυτό είναι αδύνατον εάν δεν είναι με τρόπο αηφόρο. Και έχω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη είναι η εξής. Αν δείτε την εκβιομηχάνηση με τρόπο αηφόρο, ποιους κλάδους θα βλέπατε εσείς. Και να τελειώσω, να τελειώσω κύριε Πρόεδρε. Συνάδελφοι, πρέπει να τηρήσουμε το χρόνο. 45 συνάδελφοι περιμένουν. Πρέπει λοιπόν να μείνουμε εντός του χρόνου. Με συγχωρείτε, δύο λεπτά κυρία ε, υποψήφια επιτροπέ. Αν μου επιτρέπετε. Μου επιτρέπετε, βεβαίως. Θα επαναλάβω αυτό που είπα και προηγουμένως. Από την προηγούμενη μου απάντηση επαναλαμβάνω αυτή τη φράση ότι πιστεύω ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας βάσει και της δήλωσης του κυρίου Γιούνκερ για το πακέτο επενδύσεων των 300 δισεκατομμυρίων το οποίο επεξεργάζεται και ο μελλοντικό αντιπρόεδρος ο κύριος Κατάινεν και νομίζω θα σας παρουσιάσει συγκεκριμένες προτάσεις όταν αρχίσει η εντολή του Πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να εξασφαλίσουμε την ε, ανάπτυξη με έναν τρόπο που θα είναι αηφόρος και στο κοινωνικό επίπεδο και στο επίπεδο του περιβάλλοντος και στο επίπεδο της βιομηχανικής πολιτικής. Αναφέρθηκα προηγουμένω σε μία σειρά από κέριους τομείς. Αλλά δεν θέλουμε να δώσουμε ειδική μεταχείριση σε κανένα τομέα στην Ευρώπη, κάθε άλλο. Εγώ θα αντιμετωπίσω όλους τους τομείς τους οικονομικούς στην Ευρώπη, είτε είναι χημική βιομηχανία, αυτοκινητοβιομηχανία ή κατασκευαστικός τομέας. Όλοι αυτοί οι τομείς φυσικά είναι αλληλένδετοι με άλλους ε, τομείς ε, παροχής υπηρεσιών ή παραγωγής προϊόντων. Είπα προηγουμένως λοιπόν ότι θα εργαστούμε και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό ώστε κανένας τομέας της βιομηχανίας μας να μην βρεθεί στο περιθώριο γιατί θέλουμε να εκμεταλλευτούμε το πλήρες φάσμα δυνατοτήτων στην Ευρώπη από τις βιομηχανίες οι οποίες έχουν και συμβολικό χαρακτήρα όπως είναι η χαλιβουργία μέχρι τις, ε, οικονομικού τους οικονομικούς κλάδους που δημιουργούν θέσεις, θέσεις απασχόλησης όπως είναι ο τουρισμός. Και σα υπενθυμίζω ότι ο τουρισμό είναι η τρίτη πηγή πόρων για την Ευρώπη. Πρέπει να κατανοήσουμε λοιπόν ότι για κάθε ένα από αυτού του ε, τομεί πρέπει να σχεδιάσουμε τη δράση μα ώστε να χρησιμοποιήσουμε με το καλύτερο δυνατό τι δυνατότητε που έχουμε. Ευχαριστώ κύριο Ντούντα από τη Συντηρητική και Μεταρρυθμιστική Ομάδα. Κύριε Επιτροπέ, δύο ερωτήσεις. Πρώτον, αναφέρατε στην ομιλία σας πως συχνά επικρατούν τα τοπικά συμφέροντα και ίσως επικρατούν κάποτε η διαφθορά και η γραφειοκρατία. Ενδιαφέρον αυτό γιατί νομίζω πως η διαφθορά, η προφανής είναι εύκολο να φανεί αλλά η διαφθορά δεν είναι πάντα η παρανομία καμιά φορά είναι απλά μια προνομιακή μεταχείριση που καταστρέφει το σύστημα δημοσίων προμηθειών. Οπότε η Κομισιόν θα δει το καθόλου το θέμα των δημοσίων προμηθειών και με ποιο τρόπο. Δεύτερον, είπατε πως θέλετε να ενισχύσετε την ισχύ της εσωτερικής αγοράς και αναφέρατε ως προτεραιότητα κάποιες δράσεις που θα πρέπει να ενστιαστούν στα μέτρα εκείνα τα οποία θα μας δώσουν ένα ανταγωνιστικό πλέον έκτημα πώς θα το αξιολογούσετε αυτό σε σχέση με την αρχή της εφόρου ανάπτυξης. Ευχαριστώ. Δημόσιες ε, προσλήψεις, μάλλον συγγνώμη, δημόσιες προμήθειες. Όλοι έχουμε την εμπειρία από τις δικές μας χώρες. Σε πολλούς τομείς λοιπόν έχουμε ε, προμήθειες δισεκατομμυρίων ευρώ και οι δημόσιες προμήθειες θα πρέπει να είναι και αυτές στο επίκεντρο των δράσεών μου. Την Άνοιξη εμφανίστηκε το πακέτο νομοθετικό για τις δημόσιες προμήθειες, το οποίο από τη μία πλευρά έχει σαν στόχο να ανοίξει την αγορά των δημοσίων προμηθειών σε όλες τις χώρες. Αποτελούν το 20% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ οι δημόσιες προμήθειες, αλλά μόνο 2% από αυτές τις δημόσιες προμήθειες γίνονται σε διαμεθοριακό επίπεδο. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το υπογραμμίσουμε. Δεύτερον, το θέμα είναι η πρόσβαση στους δημόσιους διαγωνισμούς για παροχή υπηρεσιών ή προϊόντων. Τρίτον, υπάρχει το θέμα το οποίο μπορώ να το ονομάσω το θέμα της διαφθοράς. Όταν λοιπόν υπάρχουν κάποιοι κανόνες οι οποίοι είναι νομότυποι αλλά διευκολύνουν πολύ περισσότερο κάποιους ε, να πάρουν αυτές τις προμήθειες από κάποιους, από κάποιους άλλους. Πρέπει να κάνουμε λοιπόν ό,τι είναι δυνατόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πάρα πολλά που πρέπει να γίνουν. Υπάρχουν διαφορά ελλείμματα στα κράτη-μέλη που πρέπει να αντιμετωπιστούν και θέλω να πω και το εξή. Κοιτάξτε. άμα έχουμε μια καλή και σύγχρονη διοίκηση με ένα σύστημα το οποίο χρησιμοποιεί όλα τα απαραίτητα σύγχρονα μέσα, ένα σύστημα όπου είναι όλα φανερά και διαφανή, αυτό μπορεί να οδηγήσει στη μείωση της διαφθοράς σχεδόν στο 0%. Είμαι σίγουρη λοιπόν ότι μια καλή δημόσια διοίκηση και η καλή κατάρτιση μπορούν να αντιμετωπίσουν τα θέματα αυτά. Κυρία Σαρανσόνα, από την ε, φιλελεύθερη ομάδα. Κυρία Χαράνσοβα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Υποψήφια Επιτροπέ. Η Κομισιόν έχει δεσμευτεί στον νόμο περί μικρών επιχειρήσεων ε, να εφαρμόσει την αρχή ε, ξεκινάμε από τις μικρές επιχειρήσεις και έτσι θα αξιολογεί τον αντίκτυπο της νέας νομοθεσίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για τους φιλελεύθερους έχει ζωτική σημασία να γίνεται σωστά αυτή η αξιολόγηση και εμείς θεωρούμε πως υπάρχει εδώ πέρα μεγάλο περιθώριο προόδου. Παραδείγματο χάρη πρέπει να συμβουλευόμαστε του ενδιαφερόμενου, αυτού που εκπροσωπούν τι μικρομεσαίε επιχειρήσει ήδη από το πρώτο σχέδιο τη αξιολόγηση αντικτύπου. Θεωρείτε πως η αρχή αυτή εφαρμόζεται επαρκώς όταν συντάσσεται νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία και δεύτερον πώς θα φροντίσετε να γίνουν σωστά αυτές ε, αξιολογήσεις για κάθε νέο νόμο που θα προτείνετε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι αυτό ένα από τα ζητήματα το οποίο πραγματικά με ενδιαφέρει. Εντάξει, πολλά ζητήματα με ενδιαφέρουν, αλλά και αυτό ιδιαίτερα. Αν αποφασίσει κανείς να στήσει μία επιχείρηση στην Ευρώπη, δεν σημαίνει πως παλεύει ε, για να την κρατήσει λόγω των διαφόρων ε, εμποδίων και οπωσδήποτε ακριβώς το προβάδισμα αυτό των μικρών επιχειρήσεων είναι κάτι το οποίο θα προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε. Ε, όπως είπα όλα τα μέσα που έχουμε αυτή τη στιγμή στην διάθεσή μας τα οποία θα καταστήσουν δυνατή την αξιολόγηση πριν εφαρμοστεί ένας νόμος οπωσδήποτε θα τα χρησιμοποιήσουμε. Μέχρι το τέλος της διαδικασίας. Δεν είναι δυνατόν, παραδείγματο χάρη, να έχουμε αξιολόγηση αυτή και να ξέρουμε πώς αυξάνεται το γραφειοκρατικό βάρος. Κάτι θα πρέπει να κάνουμε. Θα συνεργαστούμε στενά με τον κύριο Τίμερμανς, ο οποίος θα είναι προσωπικά υπεύθυνος για αυτό το θέμα. Εγώ θα καταβάλω κάθε προσπάθεια για να γίνουν πιο απλές οι διοικητικές διαδικασίες και όσον αφορά το κόστος και όσον αφορά το χρόνο. Και κάτι το οποίο αναφέρατε κι εσείς, κυρία μου, θεωρώ πως η διαδικασία διαβούλευσης πρέπει να γίνεται με όλους τους ενδιαφερομένους. Επιχειρήσεις, καταναλωτές, μικιό, οργανώσεις καταναλωτών, όλοι πρέπει να εμπλέκονται σε αυτή την διαδικασία. Ο κύριος Ντεγιόγκ από την ΚΟΕ. E. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύρια Γιανκόψκα, εδώ. Δηλώσατε πως ε, η υγεία προηγείται της αγοράς και εγώ συμφωνώ και συμφωνεί και το Κοινοβούλιο. Αλλά το Κοινοβούλιο επίσης είναι κατά του να πάει η ευθύνη για τα φάρμακα και τον ιατρικό εξοπλισμό από τη Γενική Διεύθυνση Υγείας στη Γενική Διεύθυνση Αγοράς και Βιομηχανίας. Είδαμε πως όλες οι πολιτικές ομάδες έστειλαν μία επιστολή για αυτό το θέμα. Είστε διατεθειμένοι να στείλετε κι εσείς μια τέτοια επιστολή και να πείτε ότι δεν θέλετε αυτό το χαρτοφυλάκιο και να ξαναπάει στον συνάδελφό σας. Σας ευχαριστώ η απάντησή σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ πιστεύω πως το να μπει η φαρμακοβιομηχανία στο ίδιο χαρτοφυλάκιο με την υπόλοιπη βιομηχανία είναι λογικό. Είναι μία βιομηχανία και μάλιστα είναι η μεγαλύτερη στον κόσμο. Ε, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση ο τρίτος μεγαλύτερος εξαγωγέας φαρμάκων. Και να επαναλάβω εδώ πέρα πως η υγεία και η ασφάλεια των ασθενών θα είναι πρώτη προτεραιότητα, όπως βεβαίω και η ποιότητα και η διαθεσιμότητα των φαρμάκων. Ε, ανεξαρτήτως τώρα οργανωτικών ε, λεπτομεριών, να πω πως ε, όλοι οι σχετικοί κανονισμοί οθετήθηκαν πριν από πέντε χρόνια ούτως ή άλλως ε, στη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων υπαγόταν ο κλάδος. Ε, στο ενδιάμεσο άλλαξε και τώρα επανήλθε εκεί όπου ανήκε. Να σας εγγυηθώ, όπως τα τέσσερα σημεία τα οποία ανέφερα, υγεία, ασφάλεια, ποιότητα, διαθεσιμότητα για τα φάρμακα, θα είναι οι κορυφαίες προτεραιότητες μας. Και μου και των συναδέλφων μου. Υπάρχει άλλο ένα επιχείρημα δε υπέρ, είναι ένας καινοτόμος τομέας και θεωρώ πως το συγκεκριμένο αυτό χαρτοφυλάκιο, όπως το πρότεινε ο πρόεδρος Γιούνκερ, όπου αφενός έχουμε ενιαία αγορά, αγαθά και υπηρεσίες και από την άλλη έχουμε επιχειρήσεις, βιομηχανία και καινοτομία επίσης. Νομίζω πως όλα αυτά κατατείνουν στο να ε, υπαχθούν <clears throat> όλα σε έναν, ε, στον ίδιο οργανισμό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στην αρχή του έτους το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πέρασε μια έκθεση για την βιομηχανική πολιτική με μεγάλη προτεραιότητα, με στόχο να υπάρξει μια ανανέωση της βιομηχανικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να πάρει το χαρακτήρα της αηφορίας. Χωρίς αηφορία δεν μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί στο μέλλον εσείς μέσα στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Τι θα πράξετε ώστε αυτή η άποψη να συμπεριληφθεί στη λογική του εξαμήνου. Και δεύτερο, με ποιο τρόπο θέλετε να εξασφαλίσετε τα υψηλά πρότυπα σε ό,τι αφορά την διτή επαγγελματική κατάρτιση να διατηρηθούν και πώς θα κάνετε, τι ενέργειες θα αναλάβετε για να αντιμετωπίσουμε το θέμα της ανεργίας των νέων. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Κυρία Επίτροπος, σας ευχαριστώ. Αναφέρθηκα προηγουμένως στην εναρκτήριά μου παρουσίαση στο ότι θέλω να παρουσιάσω ένα οδικό χάρτη για, το με, για τον τρόπο με τον οποίο αποσκοπούμε να οργανώσουμε, να διαρθώσουμε τη βιομηχανική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή το φάσμα των δράσεων που θέλουμε να φέρουμε σε πέρας. Στον 21ο αιώνα η βιομηχανική πολιτική θα πρέπει να είναι μια εξισορροπημένη πολιτική, μια πολιτική όπου η ανταγωνιστικότητα, ο ανταγωνισμός, η αηφόρος ανάπτυξη και η μεταμόρφωση μια οικονομία με χαμηλές εκπομπές άνθρακος θα πρέπει να ληφθούν όλα αυτά τα στοιχεία υπόψη εξάλλου. Αυτός πρέπει να είναι και ο ρόλος της καινοτομίας και επομένως το, ο δικός αυτός χάρτης θα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην καινοτομία η καινοτομία, οι τεχνολογίες εχμής, η ενεργειακή αποδοτικότητα, η καλή χρήση των πρώτων υλών, όλα αυτά είναι ουσιαστικά στοιχεία για να είναι ανταγωνιστική η ευρωπαϊκή βιομηχανία. Κατά την άποψή μου θα πρέπει να εξυγχρονίσουμε με, την, ε, τα περιφερειακά κονδύλια, με τις ε, επιδοτήσεις για τεχνολογίες εχμής, ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις του τομείς αυτής να προχωρήσουν με τα εργαλεία λοιπόν αυτά τα οποία δεν περιλαμβάνονται μονάχα στο δικό μου χαρτοφυλάκιο αλλά περιλαμβάνονται και στο χαρτοφυλάκιο του Επιτρόπου για το Περιβάλλον και αυτού που είναι αρμόδιος για την καινοτομία νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε την ανταγωνιστικότητα, συγγνώμη, μπορούμε να κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να εξασφαλίσουμε θα προωθηθεί αυτή η βιομηχανική πολιτική. Αυτό το σύστημα τώρα που είπατε για την διπλή το διπλό σύστημα κατάρτισης δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα η Κομισιόν. Νομίζω ότι είναι ένα σύστημα το οποίο έχει λειτουργήσει μέχρι στιγμής, δεν πρόκειται να το τροποποιήσει η Κομισιόν. Μας ενδιαφέρει να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες των επιχειρήσεων και προς το παρόν δεν προβλέπεται κάποια αλλαγή εδώ. Κυρία Μπορέλη, κύριος Μπορέλη. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι πηγές θέσεων απασχόλησης, είναι οι κύριες πηγές απασχόλησης και φυσικά εξαρτώνται από την ικανότητα των ε, εργοδοτών για να μπορέσει να γίνει κάτι τέτοιο. Για ένα βιοτεχνικό εργοδότη η Ευρώπη έχει μια τελείως διαφορετική εικόνα γιατί τα, τα κριτήρια κινδύνου έχουν θεσπιστεί κυρίως με την οπτική γωνία των τραπεζών ενώ οι επιχειρήσεις οι οποίες δίνουν θέσεις απασχόλησης και ανάπτυξης δεν έχουν καμία δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στις πιστώσεις γιατί είναι ιδιαίτερα περιοριστικές οι ρυθμίσεις από την πλευρά των τραπεζών που δεν έχουν κανένα τρόπο να αντιμετωπίσουν την προσθέμενη αξία που παράγουν οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν τον άνθρωπο στο κέντρο τους. Υπάρχει λοιπόν μια τεράστια απόσταση ανάμεσα στις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το τραπεζικό σύστημα και αυτό έχει πολύ αρνητικές συνέπειες για την καινοτομία που είναι ένα σημαντικό στοιχείο του χαρτοφυλακίου σας. Σας ευχαριστώ. Η κυρία ε, υποψήφια επίτροπος, σας ευχαριστώ και πάλι. Υπάρχουν τρία πράγματα που είναι πολύ ενδιαφέροντα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η πρόσβαση σε κεφάλαια και στις αγορές βέβαια και η καλύτερη ρύθμιση. Η πρόσβαση λοιπόν στα κεφάλαια όπως είπα στις αγορές και η ρύθμιση είναι οι τρεις αυτοί τομείς στους οποίους πραγματικά με ζήλο ε, θα, πάνω στους οποίους θα εργαστώ. Πρέπει να είναι ε, και το κόστος στο δυνατόν μικρότερο. Πρέπει να σας πω ότι ε, δεν λέω λόγια μόνο. Θα κάνω, μην έχετε καμία βολία, πάνω το δυνατόν για να είναι έτσι τα πράγματα. Πιστέψτε με, το εννοώ αυτό που λέω. Και σε ό,τι αφορά την χρηματοδότηση, που είπατε, κύριε Βουλευτά, εμείς θα χρησιμοποιήσουμε όλες τις μεθόδους που έχουμε στη διάθεσή μας. Θα μιλήσουμε με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, που μέχρι τώρα ήταν ε, υπεύθυνο για πολλά εργαλεία που έδωσαν σε αρκετές χώρες πολύ καλά αποτελέσματα. Όλα αυτά τα μέσα και όλες αυτές τις μεθόδους θα τις αξιοποιήσουμε ώστε η πρόσβαση ε, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να είναι ε, είναι φραγμοί αυτοί οι οποίοι πρέπει να αρθούν. Γιατί είναι προβλήματα που αντιμετωπίζουν πάντα οι επιχειρήσει. Για την καινοτομία, αν και δεν έχω χρόνο πολύ, θα πω πάντως δύο λόγια και για την καινοτομία. Η βιομηχανία. παράγει την περισσότερη καινοτομία, ανάπτυξη και απασχόληση. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις ε, είναι οι επιχείρησεις παράγουν περισσότερη ανάπτυξη, επαναλαμβάνω, και καινοτομία. Αυτή τη διαδικασία όμως πρέπει να τη στηρίξουμε από την αρχή. Όταν ξεκινά, για παράδειγμα, η συνεργασία των πανεπιστημίων με τη βιομηχανία, με τις επιχειρήσεις ή όταν έχουμε ένα πρωτότυπο το οποίο στη συνέχεια ε, βγαίνει στο εμπόριο. Πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να στηρίξουμε ίσως με υποτροφίες, χορηγήσεις, οποιοδήποτε άλλο χρηματοοικονομικό μέσο. Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε τώρα στις ε, ομάδες. Ε, Κύριο Σιένφελτ έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Υποψήφια Επίτροπε, νομίζω ότι για την οικονομική και την κοινωνική ανάπτυξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ σημαντικό να εξασφαλίσουμε την εύρυθμη λειτουργία τη εσωτερική αγορά και σε αυτό το πλαίσιο πρέπει βέβαια να εφαρμοστεί πλήρω και η οδηγία για τι υπηρεσίε. Αν όμω δυστυχώ δείτε την πρακτική, θα διαπιστώσετε ότι υπάρχουν πάρα πολλέ ε, ατέλειε. Υπάρχει ατελή εφαρμογή τη οδηγία αυτή και αυτό οφείλεται σε διάφορα προβλήματα και φραγμούς που έχουν να κάνουν με την πρόσβαση στις αγορές. Για παράδειγμα, δημόσιες προμηθείες υπάρχει βέβαια και το πρόβλημα της διαφθοράς που αναφέρθηκε και από προηγούμενους. Αν υπάρχει υπερίθμιση, αν υπάρχει γραφειοκρατία ιδίως, ιδίως για τα κλειστά επαγγέλματα. Είναι αυτά προβλήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και με όλα αυτά κατά νου λοιπόν σας ερωτώ, κύριε υποψήφια Επίτερο, πώς μπορούμε να μειώσουμε αυτά τα αρνητικά φαινόμενα. Ήξερε ίσως την ερώτηση από πριν λέει ο πρόεδρος, η κυρία και οπότε μπορεί να απαντήσει. Τι να σας κάνω, αυτή είναι η δημοκρατία, τι να σας κάνω κυρία μου λέει ο κύριος Μπούζεκ απάντηση. Ακούστε, ήδη έχω πει ότι δεν μπορεί να υπάρξει ενιαία αγορά εάν δεν ε, γίνουν αυτά που πρέπει για τις, αγαθ, για τις υπηρεσίες και τα αγαθά. Αυτό που απαιτεί η κοινή αγορά. Είπα λοιπόν ότι έχω κάποιες προτεραιότητες και η μόνο ένα προτεραιότητα σίγουρα θα είναι η οδηγία για τις υπηρεσίες που πρέπει να υλοποιηθεί. Όπως και η νέα αναθεωρημένη οδηγία για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Μηδενική θα είναι η ανοχή μας για όσους δεν εφαρμόσουν την οδηγία. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό μερίδιο της αγοράς μας. Έχουμε την οδηγία επιτόπου που ισχύει πια ε, πρέπει να εφαρμοστεί pewien raport o przeszkodach e, Σε ό,τι αφορά τώρα τα δυνητικά εμπόδια ή προβλήματα, στα μέσα του 2015 θα σας ε, παρουσιάσουμε μία έκθεση για ποια είναι τα προβλήματα τα οποία ενδεχομένω ε, παρεμποδίζουν ε, την εφαρμογή της οδηγίας. Και τώρα το δεύτερο τμήμα της ερώτησής σας για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, ποια είναι τα προβλήματα εκεί και τι γίνεται και με τα επαγγελματικά προσόντα. Όπως γνωρίζετε, έχουμε την νέα οδηγία από το 2012. Πολλές τροποποιήσεις και νέα μέτρα σε ό,τι αφορά τα επαγγελματικά προσόντα που αναγνωρίζονται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα συνεργαστώ λοιπόν με τους ενδιαφερομένους ε, φορείς, τους κλάδους αλλά και τα, ε, τους εκπροσώπους των κρατών μελών ώστε όλα τα χρήστα εμπόδια να τα εξαλείψουμε. Κυρία Ροντρίγκε. Κυρία Υποψήφια Επίτροπε, η ενία αγορά μπορεί να δημιουργήσει πολλές δυνατότητε ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων απασχόληση. Επίσης όμως μπορεί να υποσκάψει τα κοινωνικά μας πρότυπα εάν δεν υπάρξει σωστή ρυθμισή τη. Το ερώτημά μου είναι πώς θα λάβετε υπόψη την, ε, τις αρχές που περιλαμβάνονται στην ε, συνθήκη της Λισαβόνας για την συμπερίληψη και της κοινωνικής διάστασης όταν κάνετε την εξάντε ή την εξπόστ αξιολόγηση των πολιτικών. Και τέλος, ποια είναι η προσέγγιση που έχετε σε σχέση με την αρχή της καλύτερης κανονιστικής ρύθμισης. Κύριε Επίτροπος. Σας ευχαριστώ. Πιστεύω ότι η κοινωνική διάσταση στην εσωτερική αγορά έχει ένα προεξάρχοντα ρόλο. Και στην βιομηχανική πολιτική επίσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να υπάρχει. Θα πρέπει να υπάρξει μια προσέγγιση ισορροπημένη και η εσωτερική αγορά δεν είναι αυτός ο σκοπός. Είναι ένα εργαλείο για να μπορέσουν να δημιουργούν Θέσει εργασία και οικονομική μεγέθυνση. Θα πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο στου τομεί που έχουν μεγαλύτερο δυναμικό, αλλά επίση και η κοινωνική ρήτρα που αναφέρατε, η συμπερίληψη τη μνήας του περιβάλλοντο και του, των κοινωνικών στοιχείων, όλα αυτά πρέπει να περιλαμβάνονται σε όλες τις προτάσεις. Πραγματικά θα το κάνουμε αυτό στον τομέα των δημοσίων προμηθειών. Είναι και μια ευκαιρία που μας δίνεται, ώστε με αυτή τη ρήτρα να ισχύει σε όλες τις νέες διαδικασίες δημοσίων προμηθειών. Πιστεύω λοιπόν ότι η Ευρώπη μπορεί να είναι πρωτοπόρος σε ό,τι αφορά την ποιότητα των αγαθών και των υπηρεσιών της και με την ποιότητα να μην υπάρξει τώρα κάποια σύγχυση σας είπα ότι στην αρχή ότι θέλουμε μια Ευρώπη πιο κοινωνική και πιο φιλελεύθερη συγχρόνως. Μετά από την κρίση όμως θέλουμε μια Ευρώπη η οποία να είναι οικονομική, Ευρώπη αγοράς και, και κοινωνική συγχρόνως. Σας ευχαριστώ κύριε πρόεδρος. Ο κύριος Φόξ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Εδώ μπροστά σας είμαι προηγούμενη επιτροπή ξεκίνησε μια διαβούλευση για να βρει τις, τα δέκα εκείνα νομοθετήματα τα οποία επιβαρύνουν περισσότερο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μετά εξέδωσαν μια ανακοίνωση, ένα δελτίο τύπου και μίλησαν πολύ. Αλλά λίγα πράγματα έκαναν. Οπότε θα ήθελα να μου πείτε ποιο νομοθέτημα θα θέλατε εσείς να καταργήσετε για να βοηθήσετε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ένα πείτε μου. Ξέρω τον κατάλογο αυτόν, ξέρω ε, γιατί πράγμα μιλάτε. Δεν μπορώ να σας πω ένα συγκεκριμένο νομοθέτημα, αλλά σας διαβεβαιώ πως ε, μίλησα για 15 ολόκληρα λεπτά και δεν το συνηθίζω αυτό να μιλάω 15 λεπτά. Συνηθίζω να μιλάω λιγότερο και να δρώ περισσότερο. Θα ξαναδώ λοιπόν αυτό τον κατάλογο. Ξέρω τις επιχειρήσεις, ξέρω πώς ζουν γιατί ε, συνεργαζόμουν και με τον κόσμο της βιομηχανίας. Σας διαβεβαιώ λοιπόν πως δεν θα είναι κενό γράμμα ούτε θα θαυτεί σε κάποιο σιρτάρι αυτός ο κατάλογος θα μας απασχολήσει ήδη από τις πρώτες εβδομάδες, ε, προφανώς αν με εγκρίνετε για αυτή τη θέση. Και ίσως να μην είναι μόνο ένα νομοθέτημα, μπορεί να είναι δέκα, πάνω από δέκα. Σας ευχαριστώ. Κάλλας, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Υποψήφια Επίτροπε. Αναφέρατε τις δημόσιες προμήθειες ε, και το πώς ε, δεν λειτουργούν στην πραγματικότητα διασυνοριακά. Και ότι οι διασυνοριακές δημόσιες προμήθειες είναι μικρό ποσοστό του συνόλου. Ερωτώ λοιπόν συγκεκριμένα τι θα κάνετε εάν ε, γίνετε επίτροπος για να διευκολύνετε διασυνοριακές δημόσιες προμήθειες και ποια πρέπει να είναι τα επόμενα βήματα για να μειωθεί το διοικητικό άχθος ε, στις επιχειρήσεις. Και ένα άλλο σχετικό ερώτημα αναφέρατε και την απάτη και τη διαφθορά. Οι μελέτες δείχνουν πως 20 με 25% της, ε, του τιμήματος των συμβάσεων είναι η επιβάρνηση της διαφθοράς. Ο πρόεδρος... Με συγχωρείτε λέει ο πρόεδρος, τελείωσε ο χρόνος σας, παρακαλώ απαντήστε. Κοιτάξτε. Οι πιο συγκεκριμένες πράξεις έγιναν γιατί είχαμε ένα νέο πακέτο για τις δημόσιες προμήθειες που τέθει ενισχύ την Άνοιξη και πράγματι η διασυνοριακές ε, δημόσιες ε, προμήθειες είναι πολύ χαμηλές. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι γι' αυτό. Πιθανώς, ε, παραδείγματος χάρη, κάποιες διαδικασίες, κάποιοι διαγωνισμοί μάλλον αφορούν υπηρεσίες. Οι οποίες από την φύση τους είναι δύσκολο να παρασχεθούν ε, διασυνοριακά. Υπάρχουν όμως κάποιες λύσεις που μπορούν να αυξήσουν αυτό το ποσοστό. Και ελπίζω κατά τη διάρκεια της ε, αναθεώρησης θα κάνουμε να δούμε σαφώς ε, το εάν το πακέτο αυτό λειτουργεί ή όχι. Για τη δεύτερη ερώτηση... Ποια ήταν? Ναι. Παρακαλώ. Η δεύτερη ερώτηση αφορούσε το ζήτημα της διαφθοράς στις δημόσιες προμήθειες. Το ανέφερα. Η εμπειρία μου νομίζω δείχνει ξεκάθαρα πως ε, χωρίς ε, εξαιρετικά ε, μέτρα στον τομέα της καταπολέμησης της διαφθοράς μπορούμε να οργανώσουμε το σύστημα με τρόπο πιο διαφανή για να βλέπουμε πού πάνε τα λεφτά και για να μπορούν όλοι να παρακολουθούν τη διαδικασία της δαπάνης των δημοσίων κονδυλίων. Σας το λέω λοιπόν, δεν χρειάζεται καμία φοβερά κατασταλτική μέθοδος. Έχετε τον λόγο, κυρία Φόρτ. Το καλό νέο είναι ότι έχετε ξεμπερδέψει με το 1 τρίτο των ερωτήσεων. Δηλαδή το 1 τρίτο της ακρόασης έχει περάσει ήδη. Ο κύριος Σιλικιώτης είναι ο επόμενος ομιλητής από την ΚΟΕ. οι, επιχειρημα... οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τη ραχοκαλιά της οικονομίας στην Ευρώπη. Πώς θα ενισχύσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ότι όταν τα ήδη μειωμένα κονδύλια που δίνονται ε, στον προπλεσμό του 2015 δέχονται περισσότερες περικοπές δεν ακούσαμε κάτι συγκεκριμένο επίσης για την απλοποίηση των διαδικασιών πρόσβασης στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ή το πώς θα ελαχιστοποιήσετε τις επιπτώσεις από τις δεσπόζουσες θέσεις που κατέχουν στην αγορά οι μεγάλες πολυεθνικές. Επίσης μιλούμε για στήριξη της βιομηχανίας και δημιουργία νέου θέσεων εργασία, αλλά δεν ακούσαμε στήριξη είναι ιδιαίτερα του Νότου που βρίσκεται σε διαδικασία αναποβιομηχανοποίηση. Οι χώρε που βρίσκονται στο μνημόνιο βλέπουμε τι μικρομεσαίε επιχειρήσει επίση να χρεοκοπούν όπω είναι για παράδειγμα στην Κύπρο. Και ένα τελευταίο ερώτημα. Έχετε αναφερθεί για την ανάγκη τόνωση τη ανταγωνιστικότητα. Πώ θα ελοπίσετε αυτόν τον στόχο, θα συνεχίσετε την πολιτική για μείωση του κόστου, για μείωση των μισθών, για κουτσίρεμα των εργασιακών σχέσεων για να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί. Το μεγαλύτερο μέρος του χαρτοφυλακίου μου έχει να κάνει με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και με την ενιαία αγορά αγαθών και υπηρεσιών και φυσικά και το τμήμα της βιομηχανίας. Όλα αυτά έχουν σαν στόχο να διευκολύνουν την ζωή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και πρέπει να συμβάλλουν και οι τρεις πτυχές αυτές. Ξέρουμε όμως ότι δεν ζουν σε κενό αέρος οι βιομηχανίες. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι τμήμα ενός συνολικού πλαισίου επιχειρηματικότητα. Από την αρχή του επόμενου χρόνου θα σας παρουσιάσω, εάν με εγκρίνετε, ένα οδικό χάρτη για την, τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να υποστηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχείρησεις. Μπορώ να σας επαναλάβω αυτό που είπα προηγουμένως. Είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουμε την πρόσβαση στα κεφάλαια, στην ε, πρόσβαση στην αγορά, καλύτερη πληροφόρηση. Πολλές φορές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν πληροφόρηση, δεν ξέρουν σε ποιον πρέπει να απευθυνθούν. Πώς θα μπορέσουν να πάρουν ένα δάνειο. Είναι όλα αυτά λοιπόν ζητήματα τα οποία πρέπει να τα εξασφαλίσουμε για να μπορούν να έχουν τη σωστή χρηματοδότηση και φυσικά χρειάζεται και μια καλύτερη κανονιστική ρύθμιση για αυτές τις ε, μικρές επιχειρήσεις, μικρομεσαίες. Όπως είπε ε, και ο κύριος Φόξ, όλοι αυτοί οι κανόνες οι οποίοι δημιουργούν προβλήματα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να απλοποιηθούν και αυτό είναι απαραίτητο Πιστέψτε με ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρώπη έχουν προβλήματα τα οποία είναι κοινά σε μεγάλο βαθμό σε, από μία χώρα στην άλλη. Πρέπει να έχουμε μία σειρά από κοινέ πολιτικές για να μπορέσει το χρήμα αυτό το οποίο είναι σημαντικό να πάει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. τώρα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Εδώ είμαι. Κυρία Μπιενκόφσκα, είπατε και σας ευχαριστώ για αυτό ότι είστε ιδιαίτερα προσιλωμένοι στα περιβαλλοντικά ζητήματα, στην ε, βιώσιμη κατανάλωση. Ξέρετε όμως ότι το Ευρωπαϊκό Οικονομικό, η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή ομόφωνα πέρυσι γνωμοδότησε υπέρ μιας πιο βιώσιμης κατανάλωσης ε, για τη διάρκεια ζωής των προϊόντων της βιομηχανίας και για την ενημέρωση των καταναλωτών. Τώρα, υπάρχει μια προσπάθεια μείωσης της διάρκεια ζωής ε, στην Ευρώπη και θα αποκαταστήσει αυτό την ε, εμπιστοσύνη, θα αυξήσει την αποδοτικότητα των επιχειρήσεων και θα μειώσει και το οικολογικό αποτύπωμα. Ερωτώ, έχετε την πρόθεση να αναλάβετε πρωτοβουλίες ώστε η διάρκεια χρήσης των προϊόντων στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς να ενταχθεί στα βασικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. Έχετε κάποια προγράμματα, κάποια σχέδια να καταπολεμήσετε αυτή την προγραμματισμένη, προσχεδιασμένη παλαιότητα. Δηλαδή φθορά προγραμματισμένη κάποιων εξαρτημάτων των προϊόντων. Απάντηση. Ακούστε. Όλοι σας ε, γνωρίζετε ότι στη δεκαετία του 70 ένα προϊόν ε, λειτουργούσε για 20 χρόνια και σήμερα λειτουργεί μόνο 5 χρόνια. Υπάρχει ε, πρόβλημα, ε, θα το δούμε αυτό. Αν υπάρχουν αθέμητες εμπορικές πρακτικές, αυτές θα πρέπει να τις σταματήσουμε. Οι καταναλωτές πρέπει να ενημερώνονται σωστά. Αλλά θα πρέπει να φροντίσουμε να αποφύγουμε και την ε, ζημιά στον ανταγωνισμό. Πάντως συμφωνώ με αυτή σας την ανησυχία. Πρόεδρος Μάργκοτ Πάρκερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλό σας απόγευμα. Κύριε Ποσήφη Επιτροπή, μόνο η Κομισιόν μπορεί να ξεκινήσει μια διαδικασία κατάργησης ε, κανονισμού, ενώ στις γραπτές σας απαντήσεις λέτε ότι θα πρέπει να μειώσουμε την γραφειοκρατία. Πόσα νομοθετήματα, οδηγίες, κανονισμούς ε, προτείνετε εσείς να καταργηθούν ο ρόλος σας, περιλαμβάνει και τις ΜΜΕ. Ε, το άχθος ε, για, από την πολλή ρύθμιση πέφτει κυρίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν μπορούν να επομιστούν το διοικητικό κόστος οικονομιών κλίμακας, ενώ οι μεγάλες επιχειρήσεις ενθαρρύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργεί όλο και περισσότερες ρυθμίσεις και νομοθετήματα, γιατί ξέρουν ότι τους μικρούς ανταγωνιστές και τους νησερχόμενους στην αγορά τους κόβει τα πόδια. Εσείς ε, τι εμπειρίες έχετε είχατε ποτέ μια μισθωτή αμοιβόμενη απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα. Nie byłam nigdy pracownikiem prywatnego sektora, natomiast e, przez 20 e, Εργαζόμουν για 20 χρόνια ε, σε κάποια σε μέσα στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στο τι θέση, επόμενη θέση δεν είχα. Ε, ξέρω τι αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις λόγω της ε, νομοθεσίας στο εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο που δεν είναι η δέουσα. Σίγουρα υπάρχουν προβλήματα γραφειοκρατικά τα οποία δυσκολεύουν για να μην πω ότι κάποιες φορές ε, καθιστούν αδύνατο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπορέσουν να δραστηριοποιηθούν ελεύθερα. Όμως όπως είπα, στην παρούσα φάση δεν θα ήθελα και δεν μπορώ να σας πω ότι θα, βάλουμε, θα φέρουμε ένα νέο καινούργιο νομοθέτημα και θα καταργήσουμε δύο αλλά ήδη έχουν ξεκινήσει κάποιες προσπάθειες από, το, από την προηγούμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα ήθελα να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια για να δούμε ποιες είναι οι νομοθετικές πράξεις οι οποίες πρέπει να καταργηθούν. Και θα πρέπει να περιοριστεί η θέσπιση νέων στο απαραίτητο μόνο. Ευχαριστώ. Νίκολας Μπέι είναι ο επόμενος. Euh, Κυρία Πρόεδρε, σε μία απόφαση του 2012 ελήφθη μία προστατευτική ρύθμιση ένας ε, δασμός αντι-dumping εναντί προϊόντων που ερχόντουσαν από το, την Κίνα και το Βιετνάμ. Για πρώτη φορά λοιπόν υπήρξε αυτή η νυφάλια άποψη. Δεν πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίζει να έχει τους ε, εταίρους της έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση να παραβιάζουν τους κανόνες του ΠΟΕ και να προστατεύουν τις δικές τους βιομηχανίες και θέσεις εργασίας. Η Ευρώπη και οι λαοί της Ευρώπης έχουν δείξει ότι δεν πιστεύουν πια σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, τον παγκοσμιοποιητικό τρόπο αυτό που ουσιαστικά επιτρέπει την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων αλλά όχι και των ανθρώπων. Πρέπει τα κράτη μας να αποκτήσουν και πάλι την οικονομική του κυριαρχικότητα, είσαστε έτοιμοι να προχωρήσετε στην προστασία των κρατών μας και των ε, λαών μας ή θα συνεχίσετε να έχετε τις ΗΠΑ και τους άλλους παγκοσμιοποιητές να μας τραβάνε το μανίκι. Σας ευχαριστώ, λέει η πρόεδρο, λέει η κυρία Πιενκόφσκα. Πιστεύω και θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο σε αυτό το θέμα. Είπαμε ότι δεν πρέπει να αντιμετωπίζουμε δογματικά τα θέματα αυτά και θέλω να επανέλθω σε αυτή τη φράση. Μια βασική προϋπόθεση είναι η Ευρώπη να εξακολουθήσει να είναι μια ζώνη του κόσμου η οποία δημιουργεί ε, θέσεις απασχόλησης και οδηγεί σε μεγάλη ευμάρεια για τους ε, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υποστηρίξουμε την πολιτική ανταγωνισμού. Χρειαζόμαστε μια πολύπλοκη προσέγγιση. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και την βιομηχανική πολιτική, αλλά και μια ξεχωριστή πολιτική για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να θέσουμε ένα αμφιβάλλο, ένα αμφιβόλο, μια σειρά από υψηλά πρότυπα τα οποία έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, όταν μιλάμε για τη φιλελευθερωποίηση των παγκοσμίων αγορών, αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Εγώ είμαι υπερήφανη για τα υψηλά πρότυπα που έχουμε. Πρέπει λοιπόν να δράσουμε ενεργά για να προστατεύσουμε τα πρότυπα αυτά και το κεκτημένο που έχουμε με όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Και επομένως θα πρέπει στις διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του ΠΟΕ, να χρησιμοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Από την άλλη πλευρά η Ευρώπη δεν μπορεί να κλείσει τον εαυτό της και να απομονωθεί από τον υπόλοιπο πλανήτη. Υπάρχει πολύ σημαντικό ε, πολύ σημαντικές εμπορικές ροές με τρίτες χώρες και όταν πρόκειται για την καινοτομία η Ευρώπη είναι ακριβώς ο χώρος όπου γίνονται πολλά πράγματα στον τομέα της καινοτομίας. Αυτό θα πρέπει να συνεχίσει να γίνεται έτσι και στο μέλλον και αυτό δεν μπορεί να γίνει με το να κλείσουμε την οικονομία μας. Θα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρξει μια ισορροπία για το παγκόσμιο εμπόριο, να διατηρήσουμε τα πρότυπά μας αφενός, αλλά από την άλλη πλευρά η Ευρώπη να είναι ένας χώρος όπου θα μπορούν να παραμένουν επιχειρήσεις και να μην μετακινούνται. Η κυρία Ναδίν Μωράνο από το ΕΛΚ. εταιρεία Κορβιζιέ στην κλωστοϊφαντουργία βρίσκεται στην ίδια θέση με πάρα πολλές άλλες ΜΜΕ. Αύξηση τιμών ενέργεια. Πάνω από το 20% του κύκλου εργασιών είναι οι λογαριασμοί ρεύματος, δύο δις και φυσικού αερίου. Το ενεργειακό κόστος μπορεί να φτάσει από το 40% έως το 75% του κόστους παραγωγής. Επίσης, τα υφάσματα τα οποία εισάγονται περιλαμβάνουν ρήπους, όπως η νονιλφενόλη και με την ε, βιομηχανία παράγονται λίματα ε, που μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα στην, ε, στον υδροφόρο ορίζοντα αν δεν τύχουν τη σωστή επεξεργασία. Άλλο κόστο και αυτό. Έχουμε επίση το σχιστολιθικό αέριο. Θα το στηρίξετε? Θα στηρίξετε τι ΜΜΕ επίση για να μπορέσουν να εφαρμόσουν τι περιβαλλοντικέ του δεσμεύσεις και έχουμε και αυτό το επενδυτικό πρόγραμμα των 300 δις. Θα βγουν από εκεί αυτά τα κονδύλια. E, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε ε, και σας ευχαριστώ και για την ερώτηση. Πράγματι είπα πως οι τιμές στην Ευρώπη είναι από τις υψηλότερες και είναι δύσκολο έτσι να παραμείνει η ανταγωνιστική οικονομία μας. Είναι προφανές πως πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε γιατί η απόφαση για το ενεργειακό μείγμα είναι απόφαση του κάθε κράτους μέλους και όχι ευρωπαϊκή. Οπότε πρέπει να τηρήσουμε τους κανόνες που έχουν τεθεί στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά όταν μιλάμε για το ενεργειακό μείγμα του κάθε κράτους μέλους είναι δική του η απόφαση. Και οπωσδήποτε η πρόσβαση στην ενέργεια και το κόστος της ενέργειας παίζουν ρόλο κλειδί όταν μιλάμε για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Χτες ο κύριος Κανιέτε ανέφερε την ανάγκη ε, σοβαρών επενδύσεων στον τομέα αυτών και, και εγώ θα τον στηρίξω. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάθε πιθανή ε, πηγή ενέργειας να τις λάβουμε όλες υπόψη. Να αναφέρατε το σχιστολιθικό αέριο, προφανώς πρέπει να λάβουμε υπόψη και το θέμα της ασφάλειας. Και βεβαίως το θέμα αυτό θα απασχολήσει το σώμα των επιτρόπων. Όπως είπατε, πράγματι το μεγαλύτερο μέρος του κόστου της παραγωγής είναι η ενέργεια και κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Σας ευχαριστώ τρεις σύντομες ερωτήσεις. Θέλετε να βοηθήσετε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Κάτι συγκεκριμένο για το πώς θα το κάνετε όμως, δεν μας έχετε πει. Η Ευρική Κεντρική Τράπεζα δίδει χρήματα τα οποία μας περνούν από ενδιάμεσους οι οποίοι καθορίζουν τον τρόπο χρηματοδότησης. Αυτό καθυστερεί τη διαδικασία και την κάνει αναποτελεσματική. Θα αλλάξετε αυτό το σύστημα. Επίσης για το σχέδιο του επιχειρήν της Ευρώπης 2020 θα λάβετε υπόψη τις διάφορες μορφές επιχειρήσεις, θα εξασφαλίσετε ισότητα ε, ανταγωνισμού μεταξύ επιχειρήσεων οι οποίες είναι ε, συλλογικές, συνεταιριστικές ή κοινωνικού χαρακτήρα και κερδοσκοπικών επιχειρήσεων. Τέλος, τα κέντρα της έρευνας. Έχουμε εκεί την ανάγκη να έχουμε δίκτυα επιχειρήσεων για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις διαφορετικές τους αδυναμίες. Εσείς θέλετε να κάνετε δράση για να βελτιώσετε αυτή τη λύση των δικτύων επιχειρήσεων για να μπορούν να έχουν τα αποτελέσματα της έρευνας. Ευχαριστώ. Μερσή λέει η κυρία Μπιενκόφσκη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα περιφερειακά κονδύλια είναι μια πολύ σημαντική πηγή χρηματοδότηση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Από την άλλη πλευρά έχουμε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, επιπλέον το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, που μέχρι στιγμής έχει παίξει ένα σημαντικό ρόλο στο να δίνει δανειοδότηση σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Και έχουμε και το ε, κόσμο, το ε, το σχέδιο κόσμο το οποίο απευθύνεται ειδικά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όλα αυτά τα χρησιμοποιήσουμε με ενεργό τρόπο. Τώρα, όταν αναμειγνύει κανείς με αυτά τα εργαλεία, τα πράγματα δυσκολεύουν. Όλα αυτά είναι δημόσιο χρήμα και πολλές φορές μπορούν να προκύψουν πρόσθετες επιβαρύσεις. Αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε λοιπόν εμείς είναι να ασκήσουμε τη μεγαλύτερη δυνατή πίεση ώστε να αρθούν όλα αυτά τα γραφειοκρατικά εμπόδια και ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή αυτές που είναι startups και ξεκινάνε. Πρέπει να υπάρχουν εργαλεία λοιπόν τα οποία δεν δημιουργούν προβλήματα και τα οποία είναι απλοποιημένα. Γεια! για την καθυστέρηση πληρωμών τώρα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. το χρονικό διάστημα για την καταβολή των πληρωμών ε, θα περάσει από 60 μέρες σε 30 μέρες. Αυτή είναι μία από τις δράσεις που ξέρω από τη δική μου πρωτοεμπειρία ότι μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολλοί επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την καθυστέρηση αποπληρωμής των προϊόντων και των υπηρεσιών τους. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτή η λύση μπορεί να εξασφαλίσει ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα μπορέσουν να έχουν μια καλύτερη υποστήριξη. Η επανεκδομηχάνηση τη Ευρώπη, κυρία Υποψήφια Επιτροπή, θα είναι πάρα πολύ σημαντική για την αναζωογόνηση τη Ευρώπη. Το γνωρίζουμε πολύ καλά. Γνωρίζουμε ότι λιγότερο η βιομηχανία σημαίνει λιγότερε θέσει εργασία, που σημαίνει κατά βάση ότι θα αναγκαστούν οι νέοι να μεταναστεύσουν όπω ήδη συμβαίνει σε πολλέ χώρε και στην Πολωνία. Και ξέρουμε ότι και στην ε, Νότια Ευρώπη ισχύει το ίδιο πρόβλημα. Αναφέρθηκαν τα προβλήματα. Υψηλό ενεργειακό κόστο. Τετραπλάσιο στην Ευρώπη σε σχέση με τι ΗΠΑ. Είπατε στην ομιλία σας ότι θέλετε να επενδύσετε σε έναν επανεκβιομηχάνηση χάρη σε μια προσέγγιση χαμηλών εκπομπών εξαιτία του άνθρακα. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι θα είστε υπέρ του περιορισμού ε, του άνθρακα ως χρήσης ενέργειας. Δηλαδή θέλετε να περιορίσετε την εξόριξη άνθρακα και τη χρήση του καυσίμου. Απάντηση. Απλά να επαναλάβω αυτό που είπα και πριν, προσέροντας μια φράση ακόμη. Το ενεργειακό μείγμα είναι μεμονωμένη απόφαση των κρατών μελών. Το κάθε κράτος μέλος θα πάρει την απόφαση από ποια πηγή και σε ποιο βαθμό πρέπει, θέλει να χρησιμοποιήσει ένα είδος καυσίμου στο ενεργειακό του μείγμα. Φυσικά θα έχουμε και μία σύνοδο κορυφή που αποφασίσει για την κλιματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλα αυτά τα θέματα τα οποία εσείς θέσατε στι ερωτήσεις σα. Δεν μπορούμε να προεξοφλήσουμε όμως προς το παρόν ε, ή να προκαταλάβουμε τις ε, αποφάσεις και τις λύσεις σε ό,τι αφορά την κλιματική πολιτική εν γέννη. Θα ήθελα να επαναλάβω αυτό που προείπα. Είναι σαφές ότι η τιμή της ενέργειας στην Ευρώπη πρέπει να πέσει ο άνθρακας είναι ένα από τα συστατικά του ενεργειακού μείγματος και φυσικά και έχει δικαίωμα να παραμείνει. Φυσικά αυτό εξαρτάται από τις αποφάσεις που θα λάβουν τα κράτη-μέλη με την προϋπόθεση ότι θα τηρούν τους κανόνες οι οποίοι έχουν θεσπιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Ε, τώρα το λόγο έχει από τον άλλο κύριο Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε Μπιανκόφσκα, η αποτελεσματική χρήση πόρων αφορά την χρήση φυσικών πόρων από πρώτες ύλες, ε, τροφή, αέρα και νερό και είναι η βάση της αλλαγής του οικονομικού μοντέλου της Ένωσης. Ως κύρια πρωτοβουλία της στρατηγικής 2020 έχει μεγάλη σημασία για τις δουλειές και την ανάπτυξη, δημιουργεί μεγάλες οικονομικές ευκαιρίες, μειώνει το κόστος και αυξάνει την ανταγωνιστικότητα θα εξοικονομήσει πάνω από 600 δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο σύμφωνα με ε, το πακέτο της Κομισιόν. Θεωρείται λοιπόν πως η αποτελεσματική χρήση των πόρων θα πρέπει να είναι στην καρδιά της σχετικής πολιτικής της Ένωσης και πως ε, όχι μόνο πάει χέρι-χέρι με την ανταγωνιστικότητα, αλλά η μία ενισχύει την άλλη. Και συγκεκριμένα συμφωνείτε ότι χρειαζόμαστε δείκτες και στόχους για την αποτελεσματική χρήση πόρων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για την πρώτη σας ερώτηση συμφωνώ πλήρως. Θεωρώ πως ένας από τους ε, στόχους ε, της ε, πολιτικής των πόρων θα πρέπει να είναι ακριβώς να δούμε και την ασφάλεια της ε, παροχής και την ε, διαθεσιμότητα σε λογικές ε, χώρες. Και εδώ πέρα βεβαίως μιλάμε για τις διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες όσον αφορά κάποιες πρώτες ύλες κλειδιά και βεβαίως υπάρχουν και κάποια πράγματα που εξαρτώνται από μας η έρευνα και η καινοτομία όσον αφορά τις πρώτες ύλες και η αποτελεσματική χρήση πόρων. Και βεβαίως ανταγωνιστικότητα όταν μιλάμε για ανακύκλωση και διαχείριση απορρίτων και νέες αγορές. Βεβαίως αυτό σχετίζεται και με την ζωή ολόκληρη ενός προϊόντος όπως αναφέρθηκε πριν από λίγα λεπτά. Οπότε συμφωνώ πως η αποτελεσματική χρήση πόρων δεν είναι κάτι το οποίο πλήττει, αλλά είναι κάτι το οποίο ενισχύει την βιομηχανία, πράγματι. Ευχαριστώ. Και η δεύτερη ερώτηση από τον κύριο Ντένις Τεγιόγκ από την ΚΟΕ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Μπιενκόφσκα, έχω μία δεύτερη ερώτηση και ελπίζω να απαντήσετε επί της ουσίας. Και οι δύο έχουμε ως προτεραιότητα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες επιβαρύνονται από κάποιες εγκληματικές δραστηριότητες, ε, ψεύτικα τιμολόγια ε, και επίσης ε, στον τομέα του franchising όπου υπάρχουν κάποιες ιδιότυπες συμβάσεις. Μπορείτε να μου πείτε συγκεκριμένα τι θα κάνετε για αυτά τα δύο θέματα και τα δύο έχουν αναφερθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως θέματα στα οποία αναμένει μια πρωτοβουλία της ε, Κομισιόν. Συγκεκριμένα σας παρακαλώ. Σας ευχαριστώ για το ερώτημά σας. Αναφερθήκαμε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για την πολιτική στο βιομηχανικό τομέα. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις φυσικά είναι αυτέ οι οποίε παράγουν τι περισσότερες θέσεις απασχόλησης. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μα, ώστε οι αθέμητες εμπορικές πρακτικές να, να μην συνεχίσουν. Και γι' αυτό σας είχα πει πριν από λίγο ότι θα αγωνιστώ εναντίον αυτών των αθεμήτων πρακτικών σε ό,τι αφορά και την παροχή υπηρεσιών και στην ε, διαδικασία του franchising που αναφέρθηκατε προηγουμένως. Τους επόμενους μήνες θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό και να δημιουργήσουμε ένα σχέδιο το οποίο θα μπορέσει να δώσει λύσεις στα θέματα αυτά, ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη ασφάλεια για τους ε, καταναλωτές αλλά και για τους εργαζόμενους. Και τονίζω ότι η κοινωνική διάσταση θα πρέπει να διατρέχει όλες τις πτυχές της βιομηχανικής πολιτικής και της εσωτερικής αγοράς και θα αγωνιστώ γι' αυτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Μπενκόφσκα, είπατε ότι το σύστημα δημοσίων προμηθειών θα είναι μια τις ε, προτεραιότητές σας. Και αυτό είναι πολύ καλό νέο για τους φορολογούμενους και για τα δημόσια κονδύλια. Έχουμε νέα οδηγία, έχουμε νέα μέσα. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη επίσης τα κοινωνικά περιβαλλοντικά κριτήρια και η τιμή να μην είναι το μοναδικό κριτήριο ή το πιο σημαντικό τέλο πάντων. Έχω μια ερώτηση. Κύριε Μπινκόφσκα, τι θα κάνετε ώστε η πρόοδος στον τομέα της μεταρρύθμισης ε, των δημοσίων προμηθειών και συγκεκριμένα πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ε, και σεβασμό των περιβαλλοντικών κριτηρίων και των κριτηρίων για το δίκαιο εμπόριο δεν θα επηρεαστεί αρνητικά από τις διαπραγματεύσεις ε, για την ε, Συμφωνία Διατλαντικού Εμπορίου. Απάντηση. Θέλουμε να εφαρμόσουμε το πακέτο για τις δημόσιες προμήθειες. Βέβαια, ε, το πακέτο αυτό είναι κάτι το οποίο ε, έχει, το έχουμε κληρονομήσει εμείς από την προηγούμενη περίοδο. Εγώ θα προσπαθήσω όμως να εφαρμόσω τις διατάξεις τους. Έχουμε δύο ε, φαινόμενα, την ε, περιορισμένη συμμετοχή ξένων εταιριών ε, σε ό,τι αφορά τις δημόσιες προμήθειες και μικρή συμμετοχή των ΜΜΕ. Υπάρχουν βέβαια και κάποια καλά παραδείγματα, όπως αυτό της Πορτογαλίας, που έχουν εφαρμόσει σε μεγάλο βαθμό ένα ηλεκτρονικό σύστημα δημοσίων προμηθειών, οπότε και από την παριθμόν ένα ημέρα μεγάλος αριθμός των συμμετεχόντων. Αυξήθηκε σημαντικά αυτό δείχνει λοιπόν στην πράξη ότι η απλούστευση βοηθάει. Βέβαια, αυτά σχετίζονται με την ηλεκτρονική διοίκηση κτλ. Όμως έχουμε το παράδειγμα. Αν δηλαδή χρησιμοποιηθεί το e-procurement από τις χώρες σε ευρύτερη κλίμακα, τότε η συμμετοχή στους διαγωνισμούς ε, θα αυξηθεί για τις ΜΜΕ. Αυτό είναι σημαντικό. Τελευταίο ερώτημα για το πρώτο ήμιση των ερωτήσεων και πριν δώσω τη σκητάλη πάλι στον κύριο Γέρζη Μπούζεκ από την FTD, κυρία Μάρκοτ Πάρκερ. Βλέπω από το βιογραφικό σας ότι έχετε ένα μεταπτυχιακό σε δημόσια διοίκηση και οδηγεί σε αυτό σε εργασία στη δημόσια διοίκηση και έχετε διοριστεί στο παρελθόν υπουργό Υποδομών και Ανάπτυξης. Είστε γραφειοκράτης ουσιαστικά, όπως και ο Λόρδος Χιλ. Ποτέ δεν είχατε εκλεγεί και κανείς από τους συναδέλφους σας επιτρόπους θα εκλεγεί, απλώς θα εκλεγεί. Εγκριθείτε από το Κοινοβούλιο αλλά μόνο η Κομισιόν μπορεί να αλλάξει τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης αν τεθεί ενώπιον σας το θέμα της ε, κατάργησης νομοθεσίας, παραγωγής χάρη για το χρόνο εργασίας. Μπορείτε εσείς ως τεχνοκράτης, ως ε, γραφειοκράτης ε, καριέρας να μας δώσετε την διαβεβαίωση ότι θα πράξετε αυτό που θέλει το Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ. Γνωρίζω ποιο είναι ο ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων αλλά και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ξέρω ποιε είναι οι λειτουργίε του. Η πληροφορία που μου δίνεται νομίζω ότι δεν ευσταθεί. Που είχατε εσεί μάλλον δεν ευσταθεί. Υπήρξα γερουσιαστή στη χώρα μου και έχω κάποια εμπειρία σε εκλεγμένα αξιώματα. Γνωρίζω πολύ καλά ποιο είναι ο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ξέρω πόσο σημαντικό είναι το να μπορώ να συνεργάσω με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα κάνω ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό ώστε αυτή η συνεργασία όπως και των προκατόχων μου να είναι μια έντονη και ενεργή συνεργασία. Μίλησατε για το γραφειοκρατικό μου βιογραφικό όπως είπατε. Αν εγκριθώ ως επίτροπος θα είμαι η πιο μακριά από τη γραφειοκρατία επίτροπος που θα μπορούσατε να φανταστείτε. Η δημόσια διοίκηση θα πρέπει να λειτουργεί σαν μια επιχείρηση, όχι σαν μια γραφειοκρατία που είχαμε στο παρελθόν. Οποιαδήποτε δημόσια διοίκηση θα πρέπει να είναι αποτελεσματική. Όλες οι δημόσιες διοίκησεις θα πρέπει να λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Και αυτό έχω κάνει όπου έχω εργαστεί. Και σίγουρα θα τύχουν σεβασμού τα δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και όλες οι δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Κομισιόν ενώπιόν σας θα πραγματοποιηθούν και ο διάλογος μαζί σας θα είναι ένα από τα βασικά στοιχεία της εντολής μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε στον κύριο Ιβασκέβιτς. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Υποψήφια Επίτροπε. Ελέγχθησαν ήδη πάρα πολλά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. κυρίως γιατί πλήττεται ιδιαίτερα από τη γραφειοκρατία και τα διοικητικά εμπόδια, δεν λαμβάνεται υπόψη από τους πολιτικούς, παρά το γεγονός ότι όπως ξέρουμε εκείνη οι περισσότερες θέσεις εργασίας και η παραγωγή του μεγαλύτερου τμήματος του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Το αν θα αλλάξει αυτό ή όχι, αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εσά. Να έχετε υπόψη σας ότι όταν θέλετε να φιλελευθερωποιήσετε τις ε, ρυθμίσεις και να ενισχύσετε το διεθνές εμπόριο, θα έχετε πολλούς υποστηριχτές. Θα σας υποστηρίξουμε, αλλά θέλω και τη γνώμη σας για το εξή. Λέτε από τη μια μεριά θέλετε να ενισχύσετε τη βιομηχανική βάση στην Ευρώπη, από την άλλη μεριά λέτε ότι υποστηρίζετε την ε, εφαρμογή του ε, πακέτου για την ενέργεια, το οποίο ουσιαστικά θα αναγκάσει επιχειρήσεις να εγκαταλείψουν την Ευρώπη. Απάντηση. Πρώτον, συμφωνώ πλήρω ότι είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες υποφέρουν περισσότερο λόγω και της ευρωπαϊκής και της εθνικής νομοθεσίας, αυτό μπορώ να το επαναλάβω. Δεύτερον, σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας. και όλα αυτά που είπα προηγουμένως, δηλαδή η αναθεώρηση της υφιστάμενης νομοθεσίας και η αντιμετώπιση της νέας νομοθεσίας με εκθέσεις αντικτύπου και πριν και μετά και επίσης και η εξέτασή τους υπό το πρίσμα της βοήθειας που δίνουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όλα αυτά θα εφαρμοστούν. Για το δεύτερο όμως τμήμα της παρέμβασής σας δεν μπορώ να συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας, γιατί όπως είπα στην αρχή, η επαναβιομηχάνηση στην Ευρώπη και η διατήρηση υψηλών περιβαλλοντικών προτύπων δεν είναι αλληλοαποκλειόμενα στοιχεία. Μπορούν να διατηρηθούν και τα δύο. Έχουν ληφθεί ήδη αποφάσεις για το μέλλον της Ευρώπης που θα πρέπει να εμπλέκουν και το μέλλον των παιδιών μας και θα πρέπει να το σκεφτούμε αυτό. Η επαναβιομηχάνηση που θα δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης και αυτό θα δώσει ένα πλεονέκτημα στις ε, μικρομεσαίες. Οι μεγάλες βιομηχανίες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι υπηρεσίες και οι καινοτομίες και η καινοτομία είναι αλληλένδετα στοιχεία. Δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε κάποιο στοιχείο από αυτό το συνολικό πλαίσιο και όλα αυτά δεν έχουν κανένα αρνητικό αποτέλεσμα για την προστασία του περιβάλλοντος. Περιμένουμε τώρα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να συζητήσει τα θέματα αυτά τον Οκτώβριο και θα δούμε τι αποφάσεις θα ληφθούν. Ευχαριστώ πολύ την υποψήφια πίτροπο για αυτήν την απάντηση. Η κυρία Γκάλ Πέλτς έχει τώρα το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Υποψήφια Επιτροπή, σας ευχαριστώ για την εναρκτήρια ομιλία σας και κυρίως γιατί εκφράσατε δέσμευση να εργαστείτε για την εμβάθυνση της εσωτερικής αγοράς. Βλέπετε ότι είναι πολλά και μεγάλα τα εμπόδια. Ένα θέλω να σας αναφέρω εδώ μπροστά σας. Μπροστά σας είμαι. Έλεγα λοιπόν ότι ένα από τα εμπόδια προκύπτει όταν ένας πολίτης, για παράδειγμα, θέλει να πάρει από το ένα κράτο μέσα στο άλλο και να πάρει μαζί το αυτοκίνητό του. Ξεκίνησαν κάποιες διαβουλεύσεις, έγιναν κάποιες προσπάθειες, αλλά μπλοκάρισε το Συμβούλιο τα πράγματα ζητώντα να γίνει πρώτα μία μελέτη. Τι μπορεί να γίνει για να διευκολυνθούν οι καταναλωτές, να διευκολυνθούν οι επιχειρήσει. Απάντηση. Ευχαριστώ. Ίσως αυτό που θα σας πω είναι μια εμπειρία που έχετε και άλλοι πολλοί. Μιλάτε, αν κατάλαβα καλά, για την ταξινόμηση ενός αυτοκινήτου στην εσωτερική αγορά. Το έχουν αναφέρει αυτό οι πολίτες ως ε, μια από τις πιο προβληματικές πτυχές του να ζει κανείς ε, στην Ευρώπη. Δηλαδή συνεχώς ε, πρέπει να το ταξινομεί στη χώρα που, στην κάθε χώρα που πηγαίνει να διαμείνει. Και έχουμε λάβει πάρα πολλά παράπονα από τους πολίτες. Στόχος σε μια αγορά σίγουρα είναι να μειώσει τη γραφειοκρατία. Η πρόταση που έχει κατατεθεί δεν επηρεάζει το εθνικό δίκαιο, δηλαδή μπορεί οποιοδήποτε κράτος να φορολογεί τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που εισέρχονται στην επικράτεια. Για να ολοκληρώσω, θέλω να τονίσω το εξής. Αντιλαμβάνομαι ότι η οδηγία έχει ως στόχο τον εξορθολογισμό της διαδικασίας αυτής. Είναι κάτι πολύ σημαντικό για τους πολίτες μας. Γι' αυτό λοιπόν θα κάνω ό,τι μπορώ για να φτάσουμε σε συνένεση στο Συμβούλιο γιατί είναι μεταξύ των 20, των πρώτων 20 ε, προβλημάτων, ε, τουλάχιστον στα μάτια των πολιτών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Επίτροπε. Η Εύελιν Γκέπχαρτ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Κύριε Υποψήφια Επίτροπε, ήδη αναφέρθηκε πολλές φορές το θέμα των δημοσίων προμηθειών και στο πακέτο που αποφασίσαμε τον Απρίλιο 2014 περιέχονται κάποιες καινοτομίες μεταξύ των οποίων η καλύτερη εφαρμογή των κριτηρίων για το εργατικό δίκαιο και τις κοινωνικές υποθέσεις και θα πρέπει να τα λάβουν αυτά υπόψη και οι ανάδοχοι και οι υπεργολάβοι τους. Πώς θα φροντίσετε εσείς ε, οι μικρές αρχές που κάνουν αναθέσεις, δήμοι ας πούμε, ε, να χρησιμοποιούν αυτά τα κριτήρια τα οποία είναι και σημαντικά για την ανάπτυξη μιας περιφέρειας. Το άλλο θέμα ήταν η συζήτηση για την ε, οδηγία περί παραχωρήσεων και ακριβώς εκεί πέρα λέμε πως δεν θα πρέπει να υπάρξει πίεση για απελευθέρωση ή ή άλλων κοινωνικών ε, αγαθών και υπηρεσιών κοινή ωφέλεια. Τι θα κάνετε γι' αυτό. Τελείωσε ο χρόνος σας λέει ο πρόεδρος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αναφέρθηκα πράγματι στο θέμα αυτό. Είναι σημαντική αυτή η πτυχή των δημοσίων προμηθειών. Υπάρχουν κάποια μέσα με τα οποία τα κράτη-μέλη μπορούν να εφαρμόσουν ε, ρήτρε και καινοτόμες ε, και για το περιβάλλον και κοινωνικές έτσι ώστε τα κοινωνικά ζητήματα, τα ζητήματα καινοτομίας ε, έχουν ιδιαίτερο ρόλο στον τομέα των δημοσίων προμηθείων. Είναι μεγάλη ευκαιρία, ειδικά για τους μικρότερους φορείς, να μπουν τέτοιες ρήτρε ε, στους διαγωνισμούς. Και μαζί με τους ε, συναδέλφους μου θα πρέπει ακριβώς να δούμε τα θεσμικά όργανα τα οποία στόχο έχουν την ενημέρωση των επιχειρήσεων και θα οργανώσουμε μια εκστρατεία πληροφόρησης για να διαδώσουμε ακριβώς το μήνυμα. Και έτσι ακριβώς θα μεταδώσουμε τις βέλτιστες πρακτικές, θα δώσουμε νομικές συμβουλές και θα ξεκινήσει μια εκστρατεία ενημέρωσης όσον αφορά την διαχείριση του νερού. Δεν σκοπεύω να αλλάξω αυτό το οποίο συμφώνησε το Κοινοβούλιο με το Συμβούλιο. Ο συνεχής διάλογος με τους ενδιαφερόμενους και τους πολίτες που ενδιαφέρονται για τις πρωτοβουλίες αυτές θα συνεχιστεί, αλλά δεν έχουμε προγραμματίσει κάποια αλλαγή. Σας ευχαριστώ. Τον λόγο έχει ο Μπρόνσλα Πιέχα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Γιούνκερ είπε πώς θα αναλάβετε και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Φαρμακών με αρκετά μεγάλο προϋπολογισμό. Σκέφτομαι, έχετε ε, μεγάλη εμπειρία. Εγώ θεωρώ πως δεν έχετε αρκετά μεγάλη εμπειρία στον κλάδο αυτό. Μήπως έτσι δεν θα υπάρχει η σωστή ισορροπία μεταξύ πρόσβασης σε λύσεις και της βιομηχανίας. Να αναφέρω το παράδειγμα του Viagra. Ήταν αμερικανική ιδέα, αλλά είχε πάρα πολλές συνέπειες στις ε, τιμές των φαρμάκων σε ολόκληρο τον κόσμο. Τι μπορούμε να κάνουμε για να μειώσουμε ακριβώς αυτό το κενό, το χάσμα μεταξύ της φαρμακοβιομηχανίας και του πόσο πληρώνει ο πελάτης, ο ασθενής δηλαδή. Και επίσης το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων νομίζω ότι είναι οι λομπίστες τελικά αυτοί που επικρατούν. Σας ευχαριστώ. Αγαπητέ συνάδελφε, σας διαβεβαιώ πως ε, αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με τις πτυχές των φαρμακευτικών προϊόντων θα συνεχίσουν να το κάνουν και στο μέλλον εάν γίνω επίτροπος. Οπότε για να απαντήσω στο ερώτημά σας το ότι δεν έχω πείρα στο συγκεκριμένο τομέα δεν σημαίνει πως θα κάνει τη δουλειά μου πιο δύσκολη. Όπως ξέρετε πέρσι έγινα υπουργό ε, υποδομών στην Πολωνία και νομίζω καλά τα κατάφερα. Και η ζωή μου νομίζω και η επαγγελματική μου εμπειρία αποδεικνύει πως ε, δεν επηρεάζομαι από λομπίστες και σας διαβεβαιώ πως ε, τέτοιες πρακτικές θα είναι απαγορευμένες στις υπηρεσίες τις οποίες θα υποπτεύω. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Φιλίπ Ντεμπάκερ έχει το λόγο. Θα ήθελα να μείνω λίγο στο ίδιο θέμα. Ε, αναλάβατε τον έλεγχο της φαρμακοβιομηχανίας και είναι σημαντικό αυτό ότι έχουμε αυτή τη βιομηχανία δεδομένου και του ότι ο πληθυσμός γυράσκει τα ερωτήματά μου είναι συγκεκριμένα. Τι θα κάνετε για να ενισχύσετε το οικοσύστημα αυτό, γιατί δεν είναι μόνο οι μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείε, αλλά υπάρχουν και μικρομεσαίες που χρειάζονται βοήθεια στην ανάπτυξη νέων φαρμάκων ή ιατρικών συσκευών. Δεύτερον, ποια είναι κάποια από τα εμπόδια που βλέπετε εσείς για μια βιομηχανική πολιτική στον τομέα αυτών και τρίτον πολλές συζητήσεις βεβαίως γίνονται με τα κράτη-μέλη πολλές από τις καθυστερήσεις που βλέπουμε όταν έρχονται νέα φάρμακα στην αγορά είναι στο επίπεδο του κράτους μέλους. Τι μέσα έχετε για να, πιω... για να πιέσετε, για να δεχτούν την πολιτική σας και τα κράτη-μέλη που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για την φροντίδα των ασθενών. Σας ευχαριστώ για απάντηση. Για το ερώτημα αυτό Θα ήθελα να πω ότι αυτό το τομέα θα το αντιμετωπίσω όπως και τους άλλους τομείς. Είναι χρήσιμο, είναι σωστό να έχω στο χαρτοφυλάκιό μου και τον φαρμακευτικό τομέα. Η βιομηχανία πρέπει να απαρτίζει όλους αυτούς τους τομείς. Είναι ένας τομέας που έχει τεράστια <clears throat> συμμετοχή στην καινοτομία και στην έρευνα. Όλοι οι πόροι αυτοί λοιπόν οι οποίοι προέρχονται από το πρόγραμμα Ευρώπη 2020 και άλλα προγράμματα θα πρέπει να έχουν σαν ε, αποτέλεσμα η χειροτομία στον τομέα αυτό και φυσικά θυμάστε και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι πάρα πολύ σημαντικές στον τομέα αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει συμμετοχή τους οι μικρομεσαίες αυτές επιχειρήσεις είναι και οι τροφοδότες των μεγαλύτερων επιχειρήσεων στο φαρμακευτικό τομέα. Όλα αυτά τα κονδύλια λοιπόν και όλα αυτά τα μέσα θα πρέπει να είναι στη διάθεσή μας, στη διάθεση των ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων για να μπορούν να έχουν την απαραίτητη χρηματοδότηση για να προωθήσουν την καινοτομία και την έρευνα. Η πρόσβαση στις αγορές επίσης είναι σημαντική. Η τιμολόγηση των φαρμάκων είναι στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να παρέμβει καθόλου. Αν μιλάμε λοιπόν για την πρόσβαση και την ποιότητα των φαρμάκων, αυτό είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το επιζητήσουμε για να εξασφαλίσουμε και την ε, ασφάλεια των ασθενών. Σας ευχαριστούμε για την απάντηση. Το λόγο τώρα έχει η κυρία Σακοράφα. Κύριε Πρόεδρε, Κυρία Μπιανκόφσκα, ο κύριος Γιουγκέρ ανέφερε ρητά ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να υποστηριχθούν ιδιαίτερα επειδή αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας. Όμως, αφενός τα κονδύλια της νέας προγραμματικής περίοδου δεν είναι αρκετά και αφετέρου οι διαδικασίες έγκρισης και χορήγησης είναι τόσο γραφειοκρατικές ώστε στην πράξη ακυρώνουν την όποια πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για επανεκκίνηση πραγματικής οικονομίας. Η κρίση έκλεισε χιλιάδε μικρομεσαίε επιχειρήσει, κυρίω στι χώρε του Νότου, που του επιβλήθηκε το μνημόνιο, όπω στη χώρα μου την Ελλάδα. Απέτρεψε τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, ενώ οι προποθέσει χρηματοδότηση ευνοούν μόνο τι υγιεί επιχειρήσει που δεν έχουν επιτακτική ανάγκη υποστήριξη. Σα ρωτώ λοιπόν συγκεκριμένα, πρώτον, πώ σκοπεύετε να υλοποιήσετε τι εξαγγελίε του κυρίου Γιουγκέρ για περισσότερη ευελιξία στη διάθεση δημόσιων πόρων για την τόνωση των ιδιωτικών επενδύσεων. Και δεύτερον, είπατε ότι του χρόνου θα παρουσιάσετε ένα οδικό χάρτη για την απλούστευση του κανονιστικού πλαισίου. Προτίθεστε πέραν τη άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων να προβείτε στην αριστικοποίηση των προποθέσεων ώστε να καταστούν επιλέξιμε περισσότερε επιχειρήσει. Και τέλο, με ποιου τρόπου θα εξασφαλίσετε την δίκαιη κατανομή τη ενίσχυση μεταξύ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ευχαριστώ. Πέρασε ο χρόνο σα, η κυρία υποψήφια επίτροπο. Το έχουμε ήδη επαναλάβει σε διάφορες περιπτώσεις. Οι μικρές αλλά και οι μεσαίες επιχειρήσεις είναι η ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και στον τομέα των υπηρεσιών όσο και της παραγωγής αγαθών. Γι' αυτό θα πρέπει να τους αποδώσουμε μια ιδιαίτερη προσοχή. Συγχρόνως θα ήθελα να σας πω είναι πάρα πολλά τα προγράμματα τα οποία δίδουν χρήματα για τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν είναι λίγα. Μπορεί να χρησιμοποιούνται με γραφειοκρατικό τρόπο, μπορεί να τα χρησιμοποιούν τα κάτι μελη με λαθασμένο τρόπο. Υπάρχουν πολλές φορές εμπόδια για την πρόσβαση σε αυτά τα χρήματα, αλλά τα χρήματα αυτά υπάρχουν. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει χρηματοδότηση λοιπόν για τα προγράμματα αυτά και για όλα τα προγράμματα τα οποία λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια της περιφερειακής πολιτικής και των κρατών μελών και φυσικά υπάρχουν και τα εθνικά κονδύλια τα οποία δίδονται, μιλάμε για δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ. Όλα αυτά τα χρήματα λοιπόν θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες των επιχειρήσεων οι επιχειρήσεις θα χρειάζονται αυτά τα χρήματα για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν την καινοτομία και την ανάπτυξη στους τομείς όπου λειτουργούν. Επομένως, αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε είναι να εξασφαλίσουμε ότι τα μέσα του προγράμματος κόσμε θα κατευθυνθούν σωστά προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας ώστε να γίνει αυτό το οποίο είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν σωστά τα μέσα αυτά προς τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, βέβαια υπάρχει υποστήριξη στις εταιρικέ ε, συμπράξεις μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Απλώς σε πολλές περιπτώσεις πολλά κρατημέλη δεν θέλουν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα. Έριξον. Ευχαριστώ. Κούκου, λέει ο μιλητής εδώ μπροστά σας. Κύριος Πίτερ Έριξον. Υπάρχει ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα για την ανθρωπότητα ε, θέμα επιβίωσης, αν θα καταφέρουμε να κόψουμε την κλιματική αλλαγή. Ακούσαμε τον υποψήφιο που για την ενέργεια χθε. Στην ακρόασή του λοιπόν μίλησε για την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, άνθρακα, αέριο, ε, μίλησε για το πετρέλαιο και την πολύ άσχημη κατάσταση ε, που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Εσείς ε, θα συμβάλλετε στη χρήση άλλων εναλλακτικών πηγών ενέργειας για να εγκαταλείψουμε σιγά σιγά τα ορυκτά καύσιμα και να αντιμετωπίσουμε την αλλαγή του κλίματος ή πιστεύετε, ε, τι πιστεύετε πρέπει να γίνει με τον άνθρακα στην Ευρώπη. Η μείωσή του μήπως φρενάρει τελικά τη βιομηχανική ανάπτυξη, η μείωση της χρήσης του. Απάντηση. Θα ήθελα να επαναλάβω ότι η βιομηχανική πολιτική και η βιομηχάνηση δεν είναι ασύμβατη με τη βιώσιμη ανάπτυξη ή την φιλική προς το περιβάλλον ανάπτυξη. Υπάρχουν διάφορες αποφάσεις που έχουν ληφθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και επαναλαμβάνω ότι το κράτος μέλος το εκάστοτε επιλέγει τα συστατικά του ενεργειακού μείγματος αλλά θα πρέπει ταυτόχρονα να λάβει υπόψη και την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος. Άρα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πιο προηγμένες τεχνολογίες, πιο καινοτόμες τεχνολογίες αν χρησιμοποιείται πολύ άνθρακας. Θα πρέπει να γίνει επίσης ε, μεγαλύτερη επένδυση στην καινοτομία ώστε η παραγωγή ενέργειας και από αυτές τις πηγές να γίνει πιο καθαρή. Βέβαια, για μένα δεν υπάρχει ασυμβατότητα μεταξύ περιβαλλοντικής και βιομηχανικής πολιτικής, γιατί και οι δύο είναι απαραίτητες. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρία υποψήφια επίτροπε, είπατε ότι θέλετε να ακολουθήσετε μια οδό μηδενική ανοχή έναντι των παραβιάσεων για την οδηγία για τι υπηρεσίε. Σίγουρα η οδηγία αυτή έχει βοηθήσει τη δημιουργία τη εσωτερική αγορά που είναι η βάση του ευρωπαϊκού οικοδομήματο. Αλλά αυτή την, τα τελευταία χρόνια βλέπουμε όλο και περισσότερε στι χώρε μα να αναδύονται καταστάσει οι οποίε έχουν ένα διαφορετικό χαρακτήρα. Παραδείγματο χάρη το θέμα των μετακινούμενων εργαζομένων πολλές φορές σε υπεργολαβίες. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στους πολίτες αντί να τους βοηθήσει. Τι θα πρέπει να κάνει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση για να εξασφαλίσει ότι οι υπηρεσίες θα είναι προς όφελος των ατόμων και όχι προς ε, όφελος αρχών αφηρημένων. Πώς θα τροποποιήσετε λοιπόν τις οδηγίες για να μπορέσουν να ανταποκριθούν πράγματι σε αυτές τις ανάγκες και φυσικά πρέπει να, ακουστεί, να ακουστεί και η άποψη των μικρών εργοδοτών και επιχειρηματιών στα θέματα αυτά. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι δεν είναι εύκολο κάτι που δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα να το αλλάξουμε. Θα πρέπει να περιμένουμε τις εκθέσεις σε σχέση με τον πρώτο χρόνο εφαρμογής αυτής της οδηγίας και να δούμε πώς έγινε η εφαρμογή, αν καθυστέρησε για ορισμένου λόγους. Θα πρέπει να δούμε γιατί δεν εφαρμόζεται σωστά αυτή η οδηγία για τις υπηρεσίες και επαναλαμβάνω αυτό που είπα και προηγουμένως. Αυτή τη στιγμή για μένα το σύνθημά μου είναι να μην υπάρξει καμία ανοχή στην μη εφαρμογή αυτής της οδηγίας. Αν δούμε στην αγορά ότι υπάρχει θέληση, έλλειψη θέλησης εφαρμογής αυτής της οδηγίας, τότε θα πρέπει να σκεφτούμε και αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα, κάποια δυνατότητα τροποποίησης Μέχρι τότε όμως δεν μπορούμε να το πράξουμε. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μπέντσεν έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Μπινκόφς για την καλή εισαγωγική ομιλία, την ε, δέσμευση για καλύτερη πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση. Μιλήσατε για τα 2,3 δις ε, του προγράμματος COSME που βέβαια είναι πολύ μικρό ποσό σε σχέση με άλλα κονδύλια του προπολογισμού. Μιλήσατε επίσης για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που μπορούν να αξιοποιηθούν. Εγώ έχω ένα άμεσο ερώτημα σας απευθύνω. Σήμερα ε, εστιάζουμε στη δημόσια χρηματοδότηση, στην κρατική χρηματοδότηση. Θα δει η Κομισιόν πώς θα μπορούσε να διαφοροποιήσει περισσότερο τις πηγές χρηματοδότησης, αυτό το μείγμα. Δηλαδή, ταμεία, πώς θα, ε, κονδύλια, συγγνώμη, πώς συνταξιοδοτικά ταμεία ή άλλα ιδιωτικά ταμεία, πώς θα μπορούσαν ενδεχομένω να αποδεσμευτούν και να βελτιώσουν την πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση. Ευχαριστώ. E, e, σας ευχαριστώ για την ερώτηση αυτή, διότι πέραν όλων των εργαλείων τα οποία σας έχω μέχρι τώρα παριθμίσει, εσείς μιλήσατε για το πρόγραμμα COSME, είπατε μόλις 2,3 δις. Εγώ θα ήθελα να σας υπενθυμίσω όμως ε, ότι υπάρχουν και περιφερειακά ε, ταμεία, περιφερειακά κονδύλια. Στη χώρα που γνωρίζω καλύτερα έχουμε 5 δισεκατομμύρια μόνο για μία χώρα για, ε, από το Περιφερειακό Ταμείο. Και αυτά τα περιφερειακά κονδύλια δεν απευθύνονται μόνο σε ένα κομμάτι, σε ένα μέρος της Ευρώπης, ε, σε όλη την Ευρώπη απευθύνονται και αποδίδουν. Εμείς σίγουρα θα κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να βρούμε εναλλακτικέ πηγές χρηματοδότησης εκτός ε, του τραπεζικού συστήματος. Οι business angels, ε, κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου κτλ. Δηλαδή δεν θέλουμε να χρησιμοποιούνται μόνο τα κρατικά κονδύλια, αναζητούμε και άλλες πηγές χρηματοδότησης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό μπορώ να σας το δηλώσω σήμερα. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Ο κύριος Μάρτιν τώρα έχει το λόγο. Bonjour Madame la Commissaire désignée. Euh, la présidence italienne et la Commission européenne euh, veulent Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να αναζωογονήσει την αρχή του να φτάσουμε μέχρι το 2020 σε ένα μεγαλύτερο ποσοστό της μηχανικής παραγωγής, 25% το είπατε και εσείς. Θέλουμε όμως να έχουμε δίκαια εργαλεία. Πώς αυτό το στόχο θα τον πετύχετε και πώς θα τον, αν βέβαια αυτό αυτός ο θα τον κάνετε δεσμευτικό. Ποια νομικά μέσα θα ε, χρησιμοποιήσετε προς αυτό. Το θέμα είναι βέβαια να μην έχουμε ισοπαίδωση προς τα κάτω. Έχουμε μαζικές εισαγωγέ μεταποιημένων προϊόντων, στην, των οποίων η παραγωγή δεν ανταποκρίνεται στα περιβαλλοντικά, κοινωνικά, φρολικά μας ε, πρότυπα. Υπάρχει ένα dumping επομένω και αυτό ξέρετε ότι επηρεάζει και ο ΠΟΕ προβλέπει τη δυνατότητα παρέμβασης όταν είναι σημαντικές οι ζημιές ή οι απώλειες. Δεν θέλουμε λοιπόν ε, να ε, έχουμε μία επιδείνωση των πολιτικών μας. Ε, μήπως θα πρέπει να δούμε ξανά την πολιτική μας απέναντι σε χώρες εκ των συνόρων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανέφερα τη βιομηχανία και το ότι πράγματι χάνονται δουλειές εκεί πέρα. Μιλάμε για απασχόληση και προστασία της ε, βιομηχανίας. Όπως είπα, το 2015 θα παρουσιάσω έναν ε, οδικό χάρτη που θα συμπεριλαμβάνει τα διάφορα βήματα για να διασφαλίσουμε την ε, αναβιομηχάνηση της Ευρώπης. Προφανώς αυτό το 20% είναι πολύ σημαντικό στόχος για όλους μας αλλά πρέπει να θυμόμαστε τους τρόπους με τους οποίους θέλουμε να επιτύχουμε αυτούς τους ε, στόχους. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να ρίξουμε την κοινωνική προστασία. Νομίζω ότι η αποτελεσματικότερη χρήση ενέργειας και πόρων θα βοηθήσει όμως. Προφανώς οι δεξιότητες επίσης. Όλες λοιπόν αυτές οι πτυχές ε, που θα αναπτυχθούν στη συνεργασία με τον ε, Επίτροπο Απασχόλησης θα βοηθήσουν. Όλα αυτά νομίζω τα μέτρα θα βρεθούν στον οδικό χάρτη τον οποίο θα παρουσιάσουμε αρχές του 2015. Εγώ θεωρώ πως ε, η βιομηχανία είναι πάρα πολύ σημαντική και για την καινοτομία και την ενέργεια και για τις πρώτες ύλες και αυτό το δρόμο θα ακολουθήσουμε. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ε, παρακαλέσω να κοιτάξετε λίγο πίσω πάνω από το δεξί σας όμο γιατί η συμπρόεδρος μας τώρα θα σας κάνει μια ερώτηση. Κύρια Φόρντ, Βικτόρια Γκρέις Φόρντ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Καμιά φορά κάνουμε και εμείς ερωτήσεις. Μιλήσατε για το ότι θέλετε να προωθήσετε την ατζέντα της καλύτερης ρύθμισης και να είστε πιο φιλικοί προς τις επιχειρήσεις. Στο παρελθόν είχαμε προτάσεις από την Κομισιόν που δεν είχαν θετική αξιολόγηση αντικτύπου και καμιά φορά δεν είχαν καθόλου αξιολόγηση αντικτύπου. Θα μας διαβεβαιώσετε πως δεν θα ξανασυμβεί κάτι τέτοιο στο μέλλον. Και εάν εμείς ως βουλευτές δούμε πως ε, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία δεν είχατε εξετάσει ή υπάρχουν προβλήματα στην αξιολόγηση αντικτύπου ή θα είστε διατεθειμένοι να επανεξετάσετε αυτές τις ε, προτάσεις εντός κομισιών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Φοβόμουν ότι θα είναι φοβερή ερώτηση, αλλά μπορώ να σας απαντήσω ναι και ναι. <laughs> Ωραιότατα. να σας ενημερώσω πως μαζί με την ερώτηση της κυρίας ε, Συμπροέδρου ε, ε, κάπου έχασα και την Προεδρία. Λοιπόν, είστε στο τελευταίο τέταρτο λοιπόν των ερωτήσεων. Ευχαριστώ Γέζη. Από την Άλντε ο Μάικλς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία Υποψήφια Επίτροπε. Αναφέρατε τις μικρομεσαίες φαρμακευτικές επιχειρήσεις και τους περιγράψατε ως ε, υπεργολάβους αν άκουσα καλά. Υπάρχουν όμως ε, μικρομεσαίες τέτοιες επιχειρήσεις που είναι πάρα πολύ καινοτόμες και ερευνούν και συχνά λένε πως δεν μπορούν να έχουν αρκετά μεγάλη ελευθερία στην έρευνα και επιβαρύνονται από τη γραφειοκρατία και την υπερβολική ρύθμιση. Είστε διατεθειμένοι να δείτε το θέμα με ε, σοβαρή διάθεση για να αφήσετε ακριβώς κάποια ελευθερία σε αυτές τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επιπλέον τίθεται το ζήτημα πώς βλέπετε τη συμφωνία TTIP με τις ίπα. Θα κινητοποιηθείτε για να προστατεύσετε τα συμφέροντα της βιομηχανίας μας. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Νομίζω πως ε, οι φαρμακευτικές εταιρείες ε, όπως ε, και οι άλλες θα αντιμετωπιστούν με ιδιαίτερη προσοχή. Και έχετε δίκιο. Ο αριθμός των καινοτόμων μικρών επιχειρήσεων που μπορούν ε, να επιφέρουν μεγάλες αλλαγές, να καλύψουν μια νέα θεραπεία ή ένα νέο φάρμακο, νομίζω πως ε, είναι αρκετά μεγάλος. Οπότε η απάντησή μου είναι ναι, οπωσδήποτε θα προσπαθήσω να τη στηρίξω όταν μιλάμε για τη μείωση της γραφειοκρατίας, αλλά επίσης και όταν μιλάμε για την ε, καλύτερη πρόσβαση στην έρευνα. Και τη δεύτερη ερώτησή σας δεν τη θυμάμαι. Δεύτερη ερώτηση αφορά τα συμφέροντα της βιομηχανίας, ειδικά στην ε, συμφωνία TTIP. Ναι, η απάντησή μου είναι ναι και πάλι. Αλλά ε, στην αρχική μου ομιλία δεν ε, είχα χρόνο για να αναπτύξω το θέμα αλλά οπωσδήποτε ναι. Ελπίζω και με τη δική σας την στήριξη να αναλάβω αυτό το χαρτοφυλάκιο και οπωσδήποτε ένα από τα καθήκοντά μας θα είναι να προστατεύσουμε και την βιομηχανία παραδείγματο χάρη και όλες οι υπόλοιπες βιομηχανίες στο πλαίσιο της TTIP. Λέω ακόμη στο το ΕΛΚ. Ευχαριστώ. Θέλω να εξάρω την αποφασιστικότητα που έδειξε η κυρία Επίτροπος και ελπίζω ότι θα το αποδείξει και στην πράξη. Ιδίω έναντι των χωρών που έχουν ε, μεταγράψει την οδηγία για τα συστήματα πληρωμών για την καθυστέρηση των πληρωμών, αλλά δεν την εφαρμόσουμε. Στην ε, Ιταλία έχουμε χιλιάδε εταιρείε οι οποίε χρεοκοπούν λόγω καθυστέρηση πληρωμών από τι δημόσιε αρχέ. Θα ήθελα να σα ρωτήσω με ποιο τρόπο θέλετε να αντιμετωπίσετε τα προβλήματα αυτά και τι χώρε αυτέ, και αν είναι δυνατόν να βρείτε έναν τρόπο να υπάρξει μια ε, αποζημίωση από τα κονδύλια τα οποία πληρώνονται στα κράτη-μέλη. Θέλω να έρθω τώρα στην οδηγία Μπόλκενστάιν. Εγώ δεν συμφωνώ με την απάντηση που δώσατε. Το πρόβλημα δεν είναι μονάχα η, η, μεταγραφή της οδηγίας, αλλά και τις ανάγκες που υπάρχει για να τροποποιηθούν αυτές οι ρυθμίσεις για τις επιχειρήσεις. Είσαστε έτοιμοι λοιπόν να διαπραγματευτείτε με όλα τα κράτη-μέλη για το θέμα αυτό. Διακόπτεται η ομιλήτρια. Σας ευχαριστώ, λέει η κυρία Βιενκόφσκα. Υπάρχουν πολλές πληροφορίες που δείχνουν ότι η οδηγία για τις ε, υπηρεσίες έχει καταφέρει να μειώσει σημαντικά φραγμούς και γραφειοκρατικά εμπόδια για τις επιχειρήσεις και ιδίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα συνεχίσω όμως να ακούω τις απόψεις ε, όλων των βουλευτών και όλων των κρατών μελών για ενδεχόμενους φραγμούς σε σχέση με την εφαρμογή της οδηγίας αυτής. Στους επόμενους μήνες θα προσπαθήσω να επικαιροποιήσω τα στοιχεία που έχει η Κομισιόν με τελευταία έρευνα το 2012 όταν έγινε μια προσπάθεια να καταμετρηθεί ο αντίκτυπος της ε, οδηγίας για τις επιχειρήσεις. Ξέρω ότι υπάρχουν χώρες όπως είναι η Ιταλία που έχουν ήδη προσαρμόσει μια φορά την ε, ε, νομοθεσία τους και τώρα γίνονται διαπραγματεύσεις και συνομιλίες μεταξύ της Κομισιόν και της Ιταλίας για το κατά πόσο η Ιταλία πρέπει να αλλάξει και πάλι και περαιτέρω την νομοθεσία της. Και αυτό θα είναι αντικείμενο περαιτέρω διαλόγου με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με το Ιταλικό Κοινοβούλιο γιατί έχετε δίκιο, σε κάποιες χώρες θα πρέπει οι αλλαγές να γίνουν σταδιακά. Θα το αντιμετωπίσω λοιπόν εν καιρό το θέμα αυτό. Τελευταίες δέκα Ο Σέργιο Κοφεράτη από τους Σοσιαλιστές. Σας ευχαριστώ κυρία υποψήφια ε, Επίτροπε. Επανέρχομαι στο θέμα της στρατηγικής Ευρώπης 2020. Υπάρχει η πρόταση μεταρρύθμιση τη και θα ήθελα να ξέρω πώ εσεί θέλετε να συμβάλλετε σε αυτή τη μεταρρύθμιση, την αναθεώρηση, πώ θα μπορέσετε να επιφέρετε αλλαγέ οι οποίε θα ενισχύσουν την ολοκλήρωση τη εσωτερική αγορά. Στο πλαίσιο αυτό θα ήταν χρήσιμο να γνωρίζω και ποια είναι η άποψή σα για την εξωτερική διάσταση τη ευρωπαϊκή ενιαία αγορά. Πιστεύετε ότι θα θέλατε να εφαρμόσετε την αρχή τη αμοιβαιότητα εναντί τρίτων χωρών, κάτι το οποίο για μένα έχει μεγάλη σημασία, ιδίω σε ό,τι αφορά τομείς κέριους της ε, εσωτερικής αγοράς, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως. Επομένως, να υπάρξει πλήρης πρόσβαση στην αγορά και στους δημόσιους, στις δημόσιες προμήθειες και διαγωνισμούς. Να υπάρξει κυρίως μια αμοιβαιότητα με τις πιο αναπτυγμένες χώρες είναι πάρα πολύ σημαντική για μένα. Το πιστεύετε κι εσείς. Σας ευχαριστώ. Πιστεύω ότι η στρατηγική Ευρώπη 2020 θα πρέπει να αναζητήσει έναν ρόλο για την ε, εσωτερική αγορά. Μία λοιπόν από τις δικές μου ευθύνες θα είναι αυτή η πτυχή να είναι ένας πυλώνας και να στηριχθεί στο πλαίσιο του λεγόμενου Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Επίσης μπορώ να σας πω ότι θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η κοινή αγορά να είναι προτεραιότητα στο πλαίσιο της στρατηγικής 2020. Σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με τρίτες χώρες, ε, και το είπα και στην ομιλία μου νωρίτερα, η αρχή της αμοιβαιότητας, αλλά και ε, τα αμοιβαία ωφέλη, ε, η ανάγκη να, έχουμε, να αντλήσουμε αμοιβαίο στα ωφέλη, είναι οι βασικές αρχές. Άρα η αμοιβαιότητα, όπως είπατε, βέβαια πολύ σωστά θα φροντίσω να εφαρμοστεί. Σαλίνη τώρα από το ΕΛΚΑ. Μερσή. Εγώ θα ήθελα να έρθω στη Χαλιβουργία. Έχουμε μια μεγάλη πρόκληση στην Ευρώπη, η οποία αφορά τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε τη στρατηγική δυναμικότητα αυτού του τομέα, που το έχει αναγνωρίσει αυτό το γεγονός και η Κομισιόν. Αυτή τη στιγμή όμως θα πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να εξισορροπήσουμε τον αντίκτυπο της υψηλής, του υψηλού κόστους της ε, ενέργειας στην Ευρώπη με την ανάπτυξη αυτού του στρατηγικού και νευραλικού τομέα. Δεν είναι μοναχά δημιουργός ε, προσθέμενες αξίες αυτός του τομέας, αλλά και δημιουργός θέσεων απασχόλησης, είτε στην Ιταλία, είτε στη Γερμανία, είτε σε άλλες χώρες του κόσμου. Θα ήθελα λοιπόν να δω αν μπορεί να υπάρξει καμία δυνατότητα να εξισορροπήσουμε τις δύο αυτές ανάγκες και να σεβαστούμε το στρατηγικό χαρακτήρα του χαλιβουργικού τομέα και επίσης επειδή εσείς έχετε εμπειρία ως υπεύθυνοι για τα περιφερειακά ταμεία, αν θεωρείτε ότι μπορεί να χρησιμοποιηθούν περιφερειακά κονδύλια για να υποστηρίξουν αυτή την επαναβιομηχάνηση συγκεκριμένα στη Χαλιβουργία. Σας ευχαριστώ. Ο τομέας της Χαλιβουργίας απασχολεί 350.000 άτομα στην Ευρώπη. Είναι σίγουρα ένα σημαντικό κομμάτι της βιομηχανίας μας. Χάρη στον προηγούμενο επίτροπο, τον τέος επίτροπο κύριο Ταγιάννη, έχουμε πλέον αυτό το σχέδιο δράσης για, για το χάλιβα στην Ευρώπη. Ένα σχέδιο το οποίο εκπονήθηκε σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη, τους κοινωνικούς εταίρους. Συμφωνήθηκε μάλιστα και η κοινή θέση και πλέον έχει οριστεί ένας δρόμος που θα μας οδηγήσει εκτός κρίσης. Και έχουν ξεκινήσει δραστηριότητες που προβλέπει αυτό το σχέδιο. Εγώ προσωπικά θα ασκήσω πίεση στα κρατημέλη για να εφαρμόσουν όλες τις δράσεις που προβλέπονται και οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο της αρμοδιότητάς τους. Μου. Θα ήθελα να επαναλάβω ότι στην περίπτωση της χαλιβουργίας Ουσιαστικά ε, είναι ένα σύστημα συγκοινών των δοχείων, όπως βέβαια αυτό ισχύει και για άλλους κλάδους. Η στήριξη της αυτοκινητοβιομηχανίας, ε, δηλαδή ειδική ε, δράση και για το κατασκευαστικό κλάδο. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Άρα πηγές ενέργειας. Όλα αυτά, η όλοι αυτοί είναι δυνα, δυνητικά πελάτες της χαλιβουργίας, της ευρωπαϊκής χαλιβουργίας. Άρα είναι αμφίδρομο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα περιφερειακά κονδύλια, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μεγάλο μέρος αυτών των κονδυλίων ε, για τη χαλιβουργία, όπως παραδείγματος χάρη για την καινοτομία, για τη βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων, ε, την επιμόρφωση, γιατί ξέρουμε ότι στον τομέα αυτό απασχολούνται άτομα με πολύ μεγάλη δίκευση. Είναι μια δυνατότητα λοιπόν και μπορεί να γίνει αυτό. Υπάρχουν μέσα λοιπόν, αυτά θα πρέπει όλα να τα αξιοποιήσουμε από κοινού και να τα εφαρμόσουμε με συνέπεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ. Γκρίφιν τώρα από τους Σοσιαλιστές Δημοκράτες. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υποψήφια Επίτροπε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να καταπολεμήσει τις ε, κοινωνικές ε, και εδαφικές ανισότητες κατά προτεραιότητα. Η Νέα Επιτροπή θα πρέπει να φροντίσει ε, ότι η βιομηχανική πολιτική θα επιτρέψει την ανάπτυξη και στα αστικά κέντρα και στην Ήπεθρο και σε όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε καμία τοπική κοινωνία να υπολείπεται, να μένει πίσω σε τεφορά την ανάπτυξη και την απασχόληση. Όπως προείπατε, θα πρέπει η Κομισιόν με τη δράση της να ε, δώσει κοινωνική διάσταση σε όλες τις πολιτικές οικονομικής διακυβέρνησης ή την πολιτική, τη βιομηχανική. Τι μέτρα θα πάρετε ώστε να κλείσει το κενό, ε, το χάσμα που έχει να κάνει και με την υποεκπροσώπηση, την εκπροσώπηση των φίλων ή όλων των ε, ε, φιλετικών ομάδων και τι θα κάνετε για να μειώσετε τις ανισότητες ε, στον τομέα της ανάπτυξης και της απασχόλησης ε, μεταξύ των νέων, για παράδειγμα, πώς θα ωφεληθούν από την πρωτοβουλία για περισσότερες θέσεις εργασίας και ανάπτυξη. Απάντηση. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις αυτές. Θέσατε ένα ζήτημα που είναι στόχος της περιφερειακής πολιτικής. Γιατί ένας από τους στόχους της περιφερειακής πολιτικής είναι η εξάλληψη αυτών των ανισοτήτων ε, ή χάσματος που μπορεί να υπάρχει μεταξύ διαφόρων κοινοτήτων. Όπως γνωρίζετε, η περιφερειακή πολιτική ίσως να υποτιμάται σε πολλά κράτη-μέλη, όμως υπάρχει αυτή η πολιτική, σε όλα τα κράτη-μέλη ασκείται. Σίγουρα υπάρχουν αντιπληξιακά προβλήματα σε κάποιες περιφέρειες και τότε ε, μπαίνουν σε εφαρμογή τα μέτρα της περιφερειακής πολιτικής. Έχει εργαλεία η περιφερειακή πολιτική για να εξαλείψει τα κενά, τα μειονεκτήματα και υπάρχει και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο που κατά κάποιο τρόπο έχει ένα κακό όνομα στην Ευρώπη που για μένα δεν είναι λογικό, αλλά τέλος πάντων μπορούν όμως με, και με το ΕΚΤ να λυθούν αυτά τα προβλήματα, τέλος πάντων να μειωθούν και ε, το μόνο που πρέπει να γίνει είναι να χρησιμοποιηθούν σωστά όλα αυτά τα μέτρα και εργαλεία που υπάρχουν και για τη μείωση ανεργίας των θα μιλήσω με τον αρμόδιο για την Περιφερειακή Πολιτική Επίτροπο. Έχω και εγώ εμπειρία και είμαι βέβαιη ότι ε, θα μπορέσω να την αξιοποιήσω στο πεδίο αυτό. Συνεργασία με τις τοπικές αρχές, και με τις μειονότητες όμως ή τις ομάδες πληθυσμού που είναι αποκλεισμένες από τον πυρήνα της κοινωνίας. Θα προσπαθήσουμε να κινητοποιήσουμε όλα τα μέσα για να βοηθήσουμε ιδίως τους πλέον ενδεείς. Κόλιν Λάγκεν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήθελα και εγώ να θέσω ένα ερώτημα για το ότι πήγαν τα φάρμακα στο δικό σας χαρτοφυλάκιο, όλα έγιναν πολλές ερωτήσεις και νομίζω απαντήσατε. Γι' αυτό θα κάνω μια άλλη ερώτηση. Θα ήθελα να γνωρίσω ε, εγώ τον άνθρωπο ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τόσο μεγάλο ε, χαρτοφυλάκιο. Ήσασταν μικρό κοριτσάκι όταν έγινε η αλλαγή στην Πολωνία. Θα ήθελα να μάθω πώς το ζήσατε, τι ε, εμπειρίες σας έχει διδάξει και πώς θα τα μεταφέρετε όλα αυτά στις Βρυξέλλες. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Θα προσπαθήσω εγώ να χρησιμοποιήσω την εμπειρία μου μετά το 89. Αν μου επιτρέπετε να μιλήσω προσωπικά ε, η εμπειρία μου είναι πολύ ποικιλή. Πέντε χρόνια ήμουν μόνο μητέρα και μετά επέστρεψα στη δουλειά όταν μεγάλωσαν κάπως τα παιδιά μου και η επαγγελματική μου ζωή ξεκίνησε το 1994 όταν ήμουν 30 ετών και έκτοτε πράγματι ξεκίνησα από τα χαμηλά και σιγά σιγά ανέβηκα. Μπορεί να μην ήταν όλα αυτά τα αξιώματα ερετά, αλλά εν πάση περιπτώσει ό,τι έκανα το έχω κάνει μόνη μου και προφανώς ε, βεβαίως τα ζητήματα που με απασχόλησαν ήταν κυρίως ζητήματα περιφερειακής πολιτικής αλλά είναι τόσο εκτεταμένος αυτός ο τομέας ε, της ευρωπαϊκής πολιτικής που σου δίνει πραγματικά τεράστια πείρα γιατί είναι ευρύτατος. Όπως ξέρετε ε, η περιφερειακή πολιτική, ε, η περιφερειακή πολιτική χρηματοδοτεί τα πάντα από τη βιομηχανία μέχρι τις κοινωνικές πτυχές μέχρι και μειονότητες κτλ. Οπότε μπορεί να μην είμαι ειδικό, αλλά μπορώ να σας πω πως μπορώ να σχηματίσω γνώμη για κάθε πτυχή αυτής της δουλειάς και ελπίζω αν δω την ε, δικιά μου την ε, εμπειρία να μπορέσω να κινηθώ σωστά και νομίζω πως διαχειρίζομαι καλά και τους ανθρώπους. Και σας ευχαριστώ και για την ερώτηση. Δεν ήταν και από τις ευκολότερες. Μαρία Γκρακίνη, Γκραπίνη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας παρακολούθησα με μεγάλη προσοχή και είναι καλό το ότι ρωτάω τώρα γιατί έγιναν ήδη πολλές ερωτήσεις. Εγώ όμως ε, έχω δύο ερωτήσεις που θα ήθελα πραγματικά να απαντηθούν. Δεν εφαρμόστηκαν σε όλες τις χώρες όλες οι οδηγίες, π.χ. για την οδηγία για, για τον ε, χρόνο εργασία, υπάρχει ο κίνδυνο κοινωνικού dumping αν δεν εφαρμόζεται παντού με τον ίδιο τρόπο. Το άλλο ερώτημα, έχετε πράγματι ένα πολύ ενδιαφέρον χαρτοφυλάκιο, αλλά εγώ δυστυχώς δεν άκουσα τίποτα το καινούριο για μέτρα τα οποία προτείνετε. Έχετε να μας πείτε κάποια καινοτομία ίσως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοιτάξτε, στο μελλοντικό μου χαρτοφυλάκιο νομίζω το θέμα των υπηρεσιών θα είναι ένα από τα σημαντικότερα και όπως είπα θα καταβάλω κάθε λογική προσπάθεια για να δω γιατί δεν εφαρμόζεται η σχετική νομοθεσία και η σχετική οδηγία και αυτή που είπατε για τε, την κοινωνική πτυχή ε, να εφαρμοστούν σωστά. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο. Εάν τα κράτη-μέλη και το Κοινοβούλιο αποφασίσουν να υιοθετήσουν κάποια νομοθεσία, είναι απαράδεκτο να μην ε, εφαρμόζονται μετά. Βεβαίως, εντάξει, μπορεί να υπάρχουν κάποια εμπόδια, κάποια προβλήματα, τα οποία μπορεί να δούμε, αλλά όπως είπα, θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να εφαρμοστούν όλα αυτά. Το δεύτερο ερώτημα ποιο ήταν, αν μπορείτε να με βοηθήσετε. για τα έργα εκείνα τα οποία, στα οποία μέχρι στιγμής δεν είχατε κάποια εμπειρία. Κοιτάξτε, δεν έχω κανένα, κανέναν άσο στο μανίκι, αλλά όπως σας είπα θα επανέλθουμε σε αυτό το οποίο είπαμε και στην αρχή. Υπάρχουν πολλά λεφτά στην Ευρώπη, αλλά δεν χρησιμοποιούνται συχνά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Μπιενκόφσκα. Μιλήσατε για την υγεία και την ασφάλεια. Το κοινοβούλιο μας διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή ε, σε επίπεδο ισότητος με το Συμβούλιο για τα επιβατικά αυτοκίνητα που θα έχουν ένα σύστημα για κλήσεις εκτάκτου ανάγκης. Όταν λένε ορισμένοι ότι δεν χρειάζεται περισσότερη Ευρώπη, αυτό το παράδειγμα δείχνει ακριβώ το αντίθετο, ότι η ολοκλήρωση οδηγεί σε καλύτερη ρύθμιση σε ουσιώδη θέματα όπως αυτά. Τρία ερωτήματα θα είναι η δυνατότητα να υπάρχουν αυτόματες κλήσεις μια από τις προτεραιότητες της θα το ε, προωθήσετε και για άλλα αυτοκίνητα. Θα ζητήσετε από το Κοινοβούλιο να το εγκρίνει το ταχύτερο δυνατό χωρίς καθυστερήσεις και μπορείτε να εξασφαλίσετε ότι οποιασδήποτε υπηρεσίες από τρίτη, τρίτα μέρη δεν θα οδηγήσουν σε άμεση εξαίρεση των προσωπικών στοιχείων. Ε, Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω το εξής το σύστημα e-call, η ηλεκτρονική αυτή κλίση, θα είναι μια προτεραιότητα για μας. Ε, μιλάμε για ιδιωτικά οχήματα. Δεν μπορώ να σας πω για άλλες κατηγορίες οχημάτων. Είναι ένα σύστημα το οποίο μπορεί να σώσει πολλές ζωές και είναι κάτι το οποίο πρέπει να το υποστηρίξουμε. Προφανώς θα πράξουμε ό,τι γίνεται για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια ταχεία συμφωνία μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και να εφαρμοστεί το μέτρο αυτό το ταχύτερο. <clears throat> Θα πρέπει όμως να έχουμε το γεγονός ότι είναι σημαντικό το θέμα των προσωπικών στοιχείων και της διατήρησης της ε, ιδιωτικότητας. Λαμβάνοντας πάντα αυτά υπόψη, γνωρίζοντας ότι το σύστημα e-call δεν έχει σαν στόχο να ε, παρακολουθήσει στοιχεία τα οποία είναι προσωπικού χαρακτήρα. Θα προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε λοιπόν να γίνουν όλα αυτά τα απαραίτητα ώστε να, με, να εφαρμοστεί το ταχύτερο δυνατό αλλά να μην χρησιμοποιηθεί για απόκτηση προσωπικών στοιχείων. Κυρία Γκέριγκεντ Επιτροπή Γιούρη και Σοσιαλιστική Ομάδα. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Υποψηφία Επίτροπε, το ερώτημα μου από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Η νομοθεσία για τα εμπορικά σήματα. Προτείνονται 64 διαφορετικές κατεξουσιοδότηση πράξεις. Δεν το τώρα 290 τις συνθήκες για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομοθετική εξουσία βέβαια ξέρουμε ότι έχει το Κοινοβούλιο και το ε, Συμβούλιο. Τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, συμφωνεί βέβαια να γίνει αυτή η εκχώρηση εξουσίας αν θέλετε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συγκεκριμένη ε, ρύθμιση, όμως το Συμβούλιο διαφωνεί. Ποιο κριτήριο πιστεύετε εσείς ότι πρέπει να εφαρμοστεί για τις κατηξιοδότηση πράξεις για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή για τα εμπορικά σήματα. Πρέπει να ισχύει το άρθρο 290 ή όχι. Απάντηση. Ευχαριστώ. Ακούστε, πρώτα απ' όλα πιστεύω ότι η θέσπιση του συστήματος των εμπορικών σημάτων, ανταγωνιστικών εμπορικών σημάτων, προσβάσιμων εμπορικών σημάτων είναι κάτι το οποίο νομίζω χρειάζονται πάνω απ' όλα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σίγουρα μια από τις προτεραιότητές μου θα είναι να ε, υλοποιηθεί το συντομότερο δυνατό μεταρρύθμιση για τα εμπορικά σήματα. Κατάλαβα ε, αυτό που εννοείται, το γνωρίζω το θέμα και γνωρίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέλεξε το δρόμο των κατεξοδότηση πράξεων και αυτό κυρίως για να εγγυηθεί κάποια ευελιξία για να είναι δυνατή η αλλαγή κάποιων πτυχών, που δεν είναι βέβαια από τις βασικές πτυχές αυτής της ε, ρύθμισης. Γνωρίζω ότι διεξάγεται διάλογος επί του παρόντος για τα θέματα αυτά, όμως Είμαι πεπισμένη ότι στην προκειμένη περίπτωση για το θέμα αυτό που είναι τόσο σημαντικό, τα εμπορικά σήματα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα πρέπει να μας διέπει ο κοινό νους. Και πολύ σύντομα ελπίζω θα βρεθεί επικοδομητική λύση. Δεν μπορώ να σας πω ακριβώς στην παρούσα φάση ποια θα είναι η λύση βέβαια, όμως σας υπόσχομαι ότι θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια για να γίνει. Γιατί νομίζω ότι μπορεί να γίνει και γρήγορα. Απλά πρέπει να βρεθεί κοινό έδαφος μεταξύ των ε, εταίρων. Δεν έχει νόημα να παρατείνουμε το έργο, την εργασία μας πάνω σε αυτό το θέμα. Τελευταίες τρεις ερωτήσεις λέει η πρόεδρος. Ε, Ζήφκα από το ΕΛΚ και από την Επιτροπή Θεμάτων. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε ας παραμείνουμε στο θέμα της προστασίας, ε, της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, που είναι επίκαιρο δεδομένων των νέων τεχνολογιών και του πώς λειτουργούν οι επιχειρήσεις. Η αξία των επιχειρήσεων και δι' των μικρομεσαίων βασίζεται στο δυναμικό τους και βέβαια κυρίως στο ανθρώπινο δυναμικό τους. Πολλές φορές βέβαια έχει να κάνει με τα εμπορικά σήματα, τις γεωγραφικές ενδείξεις, ε, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και ούτω καθεξής. Και αυτές είναι σημαντικές επιχειρήσεις. Το ερώτημά μου είναι τι απλουστεύσεις αναμένονται στο μέλλον σε ό,τι αφορά την προστασία των, της βιομηχανικής ιδιοκτησίας των ΜΜΕ. Ευχαριστώ. Απάντηση. Όπως είπατε, σε σχέση με την πνευματική ιδιοκτησία, Υπάρχουν διάφοροι τομείς και πολλές πτυχές που είναι σε διαφορετικό επίπεδο. Το πρώτο επίπεδο είναι ε, το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας. Αυτό θα περικόψει το κόστος ε, κατά 80% σε σχέση με το ισχύον σύστημα προστασίας. Όμως, ε, δυστυχώς δεν έχουν εφαρμόσει σχετικές νομικές διατάξεις πολλές χώρες και όπως συμβαίνει και με την οδηγία για τις υπηρεσίες πρέπει αυτή η οδηγία να εφαρμοστεί στο συντομότερο δυνατό και αυτό θα είναι μέσα στις προτεραιότητές μου. Σε ό,τι αφορά τη μεταρρύθμιση των εμπορικών σημάτων, είναι κάτι που μόλις ανέκυψε. Εγώ πιστεύω ότι είμαστε πιο κοντά στο να βρούμε τη λύση από ότι μέχρι πρόσφατα, αλλά επειδή είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πρέπει πολύ γρήγορα, στους επόμενους μήνες, να κλείσει. Θα δούμε. Θα δούμε τι συγκεκριμένες λύσεις θα εφαρμοστούν για αυτό το θέμα. Πρέπει να πω ότι οι γεωγραφικές ενδείξεις είναι κάτι θετικό, δεν είναι υποχρεωτικές, δείχνουν, δείχνουν όμως την προέλευση ενός προϊόντος και νομίζω ότι τα σχετικά θα τα εκτιμήσουν και οι περιφέρειες της Ευρώπης. Πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με τον ίδιο ρυθμό. Τέλος, το απόρριτο των συμφωνιών, η εχεμήθεια, είναι πολύ σημαντική. Και για τις, ε, για τις ευρεσιτεχνίες ε, θα κάνω ό,τι μπορώ. Κυρία Βίλμοτ, από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Σοσιαλιστική Ομάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι εισηγήτρια για, τις ιατρικές, για τον ιατρικό εξοπλισμό και τις κλινικές δοκιμές και τα δύο έχουν μεγάλη σημασία για τη ζωή των ε, ασθενών. Στο παρελθόν ασχολήθηκα για το θέμα αυτό στην Επιτροπή Υποστασίας των Καταναλωτών και Υγείας. Δυστυχώς ο κ. Γιούνκερ θεωρεί ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν αυτά στην Επιτροπή Βιομηχανίας και στη Γενική Διεύθυνση επιχειρηματικότητας. Δίνει ένα λαθασμένο μήνυμα. Ο ιατρικός εξοπλισμός και οι κλινικές μελέτες δεν είναι για κερδοσκοπία, είναι για την υγεία των ασθενών. Θα πρέπει η διαφάνεια να είναι η προτεραιότητά μας εκεί, γιατί αυτό εξασφαλίζει την ασφάλεια των ασθενών. Είσαστε δεσμευμένοι να αγωνιστείτε για τη διαφάνεια, γιατί οι αρμόδιες γενικές διευθύνσεις θα προσπαθήσουν να αποδυναμώσουν αυτές τις ε, ε Μετά το σκάνδαλο για τα ένθετα στήθους και άλλα σκάνδαλα. Μήπως θεωρείτε ότι δεν είσαστε οι πιο κατάλληλοι για να εποπτεύετε τα θέματα αυτά και να, θα είναι καλύτερα να είναι στο χαρτοφυλάκιο του, του Επιτρόπου που ασχολείται με τα θέματα υγείας. Ευχαριστώ. Όταν πρόκειται για το πρώτο μέρος της ερωτήσεώς σας, ναι, η διαφάνεια για τις κλινικές δοκιμασίες είναι κάτι το οποίο το ζητεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η πρωτοβουλία για τα ιατρικά προϊόντα, τα φαρμακευτικά και ιατρικά προϊόντα είναι πάρα πολύ σημαντική. Πρέπει να δείτε όμως και την άλλη πλευρά, δηλαδή το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας όταν πρόκειται για δυνητική ε, καταχρηστική μεταχείριση των δεδομένων. Ο νέος κανονισμός για τις κλινικές δοκιμασίες εξασφαλίζει την ισορροπία μεταξύ ανάγκης να προωθήσουμε τις κλινικές δοκιμασίες αφενός και δεύτερον να έχουμε το υψηλότερο δυνατό επίπεδο σε ό,τι αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την αξιοπιστία των δεδομένων. Θα συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη καθώς και με τον Ευρωπαϊκό Φορέα για τα Φαρμακευτικά Προϊόντα, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι όλοι οι κανονισμοί οι οποίοι εγκρίνονται έχουν υπόψη τους την ανάγκη αυτής της ισορροπίας. Σε ό,τι αφορά τώρα σε, στον ιατρικό εξοπλισμό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι υπηρεσίες της αναλύουν την κατάσταση και για τα, τα προσθετικά στήθους και έχουν αποφασίσει οι υπηρεσίες ότι σε περίπτωση ιατρικού εξοπλισμού δεν θα εφαρμόζονται οι ίδιοι κανόνες όπως για τα φαρμακευτικά συσκευάσματα. Αλλά υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για την ανάγκη να υπάρχει έλεγχος και στην παραγωγή. Όλες αυτές λοιπόν οι συστάσεις μπορεί να οδηγήσουν και σε παρέμβαση στην ίδια την παραγωγική διαδικασία. Τελευταία ομιλήτρια, η Ρόζα Εστάρα Φεραγκούτ από την Επιτροπή Μεταφορών του ΕΛΚ. Σε ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η ερώτησή μου αφορά τον τουρισμό Ξέρετε ότι η Ευρώπη είναι ο βασικός, ο, ο κυριότερος τουριστικός προορισμός. 10 εκατομμύρια ε, θέσεις εργασίας ε, ε, προσφέρει ο τουρισμός. Θέλουμε να παραμείνουμε σε ηγετική θέση. Αυτό λοιπόν σημαίνει τώρα που έχουμε με τις συνέχεια της Αβώνας αρμοδιότητες. Πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε διάφορες προκλήσεις στον τομέα του τουρισμού με πρώτη την ποιότητα. Πρώτη πρόκληση. Στην προηγούμενη νομοθετική περίοδο εγκρίθηκε μια έκθεση για την Ευρώπη για τον πρώτο τουριστικό προορισμό στον κόσμο και εκεί είπαμε ότι καλό θα ήταν να υπάρξει μια εναρμόνιση ε, στην ποιοτική αξιολόγηση ξενοδοχείων κτλ. ώστε η μάρκα, το σήμα ποιότητα να είναι εμβληματικό και εναρμονισμένο, αναγνωρισμένο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεύτερη πρόκληση η προσβασιμότητα, δηλαδή να είναι προσβάσιμος ο τουρισμός σε όλους, για τους ε, ανθρώπους με αναπηρία, για ευπαθείς ομάδες, για ηλικιωμένους και πάλι εδώ να, να κατά κάποιο τρόπο τους δείκτες προσβασιμότητας στον ε, τουριστικό κόσμο. Άλλο σημαντικό θέμα, εκπαίδευση, κατάρτιση και το να μην υπάρχει εποχικότητα, να εφαρμοστούν νέες τεχνολογίες και να υπάρχει και συνδεσιμότητα. Αυτά ευχαριστώ. Bardzo dziękuję za to pytanie, ponieważ... Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Σκοπίμως ανέφερα τον τουρισμό σε έναν από τους τομείς που θα μας απασχολήσουν. Όπως είπατε όμως, η Ευρώπη είναι ο μεγαλύτερος ε, τουριστικός προορισμός στον κόσμο. Οι μισοί ε, άνθρωποι που ταξιδεύουν έρχονται στην Ευρώπη. Σίγουρα αυτό απαιτεί την προσοχή μας. Βέβαια δεν σημαίνει ότι πρέπει μόνο στο ευρωπαϊκό επίπεδο να λαμβάνονται αποφάσεις. Παραδείγματος χάρη, ταξινόμηση των ξενοδοχείων ε, ε γίνεται σε εθνικό επίπεδο τις περισσότερες φορές, για να μην πω και σε περιφερειακό. Σίγουρα μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Για παράδειγμα, τουριστικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζονται όπως οποιαδήποτε άλλη μικρομεσαία επιχείρηση στα θέματα καινοτομία, επενδύσεων, κατάρτισης, βελτίωσης δεξιοτήτων, επιχειρηματικών δεξιοτήτων κτλ. και επομένως είναι στο πακέτο για τις ΜΜΕ. Εγώ από τη δική μου πλευρά μπορώ να δηλώσω ότι θα ξεκινήσω διαβουλεύσεις με όλους τους ενδιαφερομένους φορείς, ούτως ώστε αν είναι δυνατόν να καταρτήσουμε ένα είδος προγράμματος ή στρατηγικής για τον τουρισμό στην Ευρώπη, έχοντας βέβαια πάντα κατά νου τις επιφυλάξεις που ανέφερα στην αρχή ότι δηλαδή οι μείζονες αποφάσεις λαμβάνονται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. Δεν θέλουμε να παρέμβουμε εμείς, απλά επειδή ο τομέας αυτό είναι τόσο σημαντικός για την Ευρώπη και απασχολεί τόσα άτομα, Ίσως θα μπορούσαν να αναλυφθούν κάποιες κοινέ ενέργειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επιλεκτικές, επιλεκτικές δράσεις. Δεν θέλουμε να εθετήσουμε νέους ε, κανονισμούς για τον τουρισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ίσως όμως θα μπορούσαμε και ήδη και από αυτό το μήνα να αναλάβουμε κάποια δράση στο πλαίσιο του Υπουργικού Συμβουλίου επί Ιταλικής Προεδρίας και εκεί μπορούμε να